Για Ο τρίτος διάλογος, ε, τριμμένος διάλογος για την αναθεώρηση των κανονισμών BRD και SRM έγινε στις 26 Σεπτεμβρίου και ασχολήθηκε μεταξύ άλλων για τις ε, προϋποθέσεις χρέους, τις, ε, των structure notes, την, ε, τα cooperative groups και το αποτέλεσμα των τεχνικών εργασιών. Για τα structure notes και την ε, μεταχείριση των cooperative groups, η Κομισιόν δέχτηκε να συντάξει συμβαστικές προτάσεις που θα ε, εξεταστούν σε τεχνικές συνεδριάσεις πριν ξανασυζητηθούν σε επόμενες ε, συνεδριάσεις του τριμερούς διαλόγου. Και τώρα πάμε στα σημεία 4, 5 και 6 της μερισίας διάταξης. Έχουμε τον κύριο Κάρας, η κυρία Περβόνς Μπέρες ε, έρχεται από την Ολομέλεια, μόλις τελείωσε. Νάτι κατέφθασε πάνω στην ώρα. Ότμαρ. Ή Πενβόνς θέλει να ξεκινήσει. Ποιος από τους δυο σας. Ότμαρ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, Βρισκόμαστε στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων μετά την πρόταση και την ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης από τον Ζαν Κλοντ Γιούγκερ. Ο στόχος μου είναι η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή των Ευρωπαϊκών Αγορών να διέπεται από διαφάνεια και να επιτευχθούν συγκλήσεις. Και είναι λοιπόν κοινό μας στόχος ε, να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα και την ε, διαφάνεια στις ευρωπαϊκές αγορές, να ενισχύσουμε τη σύγκληση ε, των ευρωπαϊκών αγορών. Αυτό βέβαια πρέπει και οφείλει να γίνει μόνο μετά από κοινή προσπάθεια. Και χρειάζεται να αναγνωρίσουμε τις ε, ανισορροπίες που υπάρχουν στην δομή της. Το ζητούμενο εδώ είναι σε κάθε επίπεδο να βελτιωθεί η δομή έτσι ώστε να οδηγηθούμε το γρηγόρτερο δυνατόν στον ε, στόχο. Ο φάκελος τον οποίο ε, ξεκίνησε να δουλεύει ο συνάδελφος ε, Μπάλτς. Έχει έλθει λοιπόν σε αυτό το στάδιο. Βρισκόμαστε στις ε, προτά... τρεις προτάσεις της Επιτροπής. Έχουν κατατεθεί εκατοντάδες τροπολογίες, 1017 τροπολογίες. Και η συνεισηγήτριά μου και εγώ προτείνουμε λοιπόν τις 306 τροπολογίες να τις χωρίσουμε σε τρεις ε, κατηγορίες. Οι τροπολογίες εκείνες που αφορούν το πρώτο κομμάτι της έκθεσης ε, Είναι τροπολογίες τις οποίες ε, δεν έχουμε καταφέρει να συμφωνήσουμε. Μετά υπάρχουν οι τροπολογίες οι οποίες είναι αποτέλεσμα συμβιβασμού και από θα αποτελέσουν όχι ε, το σχέδιο έκθεσης, αλλά μια βάση για να οικοδομήσουμε την έκθεση στη συνέχεια. Ε, πρέπει, λοιπόν, να δημιουργηθεί σε διεθνές επίπεδο ε, μια ισχυρή εποπτική αρχή. Οι τροπολογίες λοιπόν της πρώτης ομάδας αφορούν αυτό. Η δεύτερη ομάδα τροπολογιών αφορά τροπολογίες στο σχέδιο έκθεσης που ε, προτείνουν τροποποίησεις. Για παράδειγμα, ε, στρατηγική εποπτική αρχή αφορά το outsourcing, τις αντιπροσωπείες, την ε, ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών ανάμεσα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η τρίτη κατηγορία τώρα αφορά τις τροπολογίες για μας οι οποίες έχουν κατατεθεί και δεν αφορούν κατά ανάγκη το ίδιο το σχέδιο έκθεσης και είναι τροπολογίες τις οποίες δεν έχουμε καταφέρει να οδηγηθούμε σε κάποια συμφωνία. Μετά, ε, για παράδειγμα, ζητήματα διακυβέρνησης, άμεσες αρμοδιότητες της ΕΣΜΑ, ε, διάφοροι παράγοντες βιωσιμότητας, κίνδυνοι, ε, no action, το ποσοστό χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα. Όλα αυτά τα ζητήματα βέβαια δεν πρέπει να χωρίσουν τους ε, δύο συνεισηγητές. Αυτή τη στιγμή, το τονίζω, είμαστε μέσα σε στάδιο επεξεργασίας όπου προσπαθούμε να βρούμε συμβιβαστικές λύσεις οι οποίες ε, θα ε, συμπεριλαμβάνουν τις ε, επιθυμίες και τις απόψεις όλων των πολιτικών ομάδων. Ε, σίγουρα δεν θα καταφέρουμε να συμφωνήσουμε σε όλα τα επίπεδα, όμως θεωρώ ότι με την διάθεση για συμβιβασμό και με την ανάλογη πολιτική βούληση θα καταφέρουμε να οδηγηθούμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Διότι μην ξεχνάτε, όσο πιο ενωμένοι είμαστε, όσο πιο ισχυροί, τόσο καλύτερα θα παρουσιάσουμε τις θέσεις μας στις ε, διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Ε, επίσης, ε, να μην ξεχνάμε τα ζητήματα της αναλογικότητας. Στον στρατηγικό σχεδιασμό επιθυμούμε και οι εθνικές αρχές να συμμετέχουν και να έχουν άποψη. Το ΕΛΚ επίσης επιθυμεί να διατηρηθεί η εθνική διάσταση στην διασυνοριακή ε, εποπτεία, ιδιαίτερα στην περίπτωση συστημικών κινδύνων. Ε, σίγουρα επιθυμεί βελτίωση του συντονισμού, πιο αποτελεσματική διακυβέρνηση και λήψη αποφάσεων χωρίς ε, περιττή γραφειοκρατία αποφυγή σύγκρουση συμφερόντων με την νομισματική πολιτική περισσότερη διαφάνεια, δυνατότητα χρονοδιαγράμματος ε, στη χρήση της ε, λύσης των δύο σταδίων, βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μην θυσιάσουμε την βιωσιμότητα στο βωμό άλλων προτεραιοτήτων. Αυτά λοιπόν εν ολίγης για τις τρεις κατηγορίες τροπολογιών Ελπίζω με βάση αυτές τις τρεις κατηγορίες να μπορέσουμε να δουλέψουμε έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε ικανοποιητικές συμβιβαστικές λύσεις. Ε, με την συνεισηγήτρια έχουμε συζητήσει σε πρώτο στάδιο, αλλά θα ήθελα εδώ να παρακαλέσω όλους τους κοιόδες ηγητές και όλους ε, εσάς τους συναδέλφους να συμμετάσχετε ενεργά στην διαδικασία. Σας ευχαριστώ. Thank you. ευχαριστώ τώρα η συνεισηγήτρια Περδόνς Μπερές. Ευχαριστώ, συνάδελφε. Παιδιά. Με μεγάλη χαρά συνεργάστηκα με τον κύριο Μπάλς ε, και θα, θα, μου λείψει τώρα που θα φύγει, γιατί ξέρετε βρίσκω χαρά στην εργασία Χαίρομαι που συνεργάστηκα με τον κύριο Καράς. Έχουμε μια ιστορία ας πούμε, συνεργασίας και ελπίζω να συνεργαστούμε καλά για να υλοποιήσουμε τον κοινό μας στόχο. Νομίζω ότι μας ενδιαφέρει όλους αυτό το θέμα. Υπό την ευρία έννοια, δηλαδή στα πλαίσια της διαπραγματευτικής ομάδας, που ώστε να καταλήξουμε εμπρόθεσμα ή περίπου εμπρόθεσμα, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε την αθεωρήση αυτών των εποπτικών αρχών πριν το τέλος της ε, εντολής και να μπούμε σε διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο. Ε, παρότι δεν ελέγχουμε εμείς την ατζέντα του Συμβουλίου, αλλά όλοι ξέρουν πολύ καλά και ο κύριος Καράς ε, στην ομιλία του υπενθύμησε τι είπε ο κύριος Γιούγκερ στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης και πόσο σημαντική είναι αυτή η μεταρρύθμιση και πόσο σημαντικό είναι να τελειώσει εμπρόθεσμα πριν το τέλος της, ε, αυτής της κοινοβουλευτικής θητείας. Για τις τροπολογίε που κατατέθηκαν υπάρχει ένας μεγάλος πλούτος, μια μεγάλη ποικιλομορφία και επιβεβαιώνονται τα διάφορα σημεία που μαζί με τον Νότμα καρά εντοπίσαμε ω σημεία διαφωνίας και επί των οποίων θα πρέπει να βρούμε μια κοινή θέση. Επίση, βλέπω την επιβεβαίωση κάποιων συμπληρωματικών στοιχείων επί των οποίων εγώ συνεισέφερα προσωπικά, ε, το να λάβουμε δηλαδή υπόψη κριτήρια για τη βιώσιμη ανάπτυξη ή το θέμα της προστασίας των καταναλωτών ως σημείο εγκάρσιο που διαπερνάει όλα αυτά τα νομοθετήματα. Υπάρχουν θέματα, επίσης, τα οποία δεν εφήγησαν από τους συνεισηγητές, ε, από τον κύριο Μπάλτς και από μένα, στην αρχική εκδοχή, και που αξίζουν όμως να τα δούμε περαιτέρω. Εν παρόδο θα αναφέρω δύο. Πρώτον, πώς εξοπλίζουμε την ΕΣΜΑ, την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, ούτω ώστε να λάβουμε υπόψη μα τα όσα ψηφίσαμε στην ε, έκθεση τη Ντανούτα Χου Χουμπνερ για τη μελλοντική εποπτεία, εάν ε, καταλήξουμε σε αυτή τη θητεία, είναι σημαντικό να ενσωματωθεί ε, στις αρμοδιότητες της ΕΣΜΑ, αυτής της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών Εφεξής ΕΣΜΑ. Το ίδιο ερώτημα θα τεθεί για τα trading venues, τους, τους, ε, τις πλατφόρμες διαπραγμάτευσης, επί των οποίων κατέθεσα διάφορες τροπολογίες. Υπάρχει ένα νέο στοιχείο, α, από τη στιγμή που κατέθηκαν τροπολογίες, ότι δηλαδή η διαπραγματευτική ομάδα θα πρέπει να λάβει υπόψη το εξή. ότι η Κομισιόν το Σεπτέμβριο δεν απέστειλε την πρότασή της ακριβώς, αλλά πήρε την πρωτοβουλία να τροποποιήσει τη δική της πρόταση. Δηλαδή, ενώ είχαμε λάβει ένα κείμενο ήδη, αυτό το κείμενο τροποποιήθηκε καθοδόν με πρωτοβουλία της ίδιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να λάβει υπόψη κάποιες εξελίξεις και την ανάγκη να παρέμβει για να ενισχύσουμε την εξουσία των εποπτικών αρχών στον ε, τομέα της ε, καταπολέμησης ε, του ξεπλήματος του χρήματος. Θα πρέπει να δούμε πώς θα παντρέψουμε όλα αυτά τα στοιχεία, θα καλύψουμε αυτές τις ανησυχίες. Εγώ, συνεισηγήτρια, ε, έχω καταθέσει σχετικές τροπολογίες, γιατί νομίζω ότι ο ρόλος αυτών των αρχών στην καταπολέμηση του ξεπλήματος είναι σαφής. Υπάρχει ένα νέο στοιχείο το οποίο έχει μπει σε πάρα πολλές τροπολογίες και επί του οποίου ομολογώ ότι έχω τις αμφιβολίες μου και μπορώ να συζητήσω το θέμα αυτό με τους συναδέλφους. Είναι το θέμα Το no action letter, σε πολύ καλά γαλλικά λέει η το είπε αγγλικά. Είναι μια διαδικασία που υπάρχει στι ΗΠΑ που επιτρέπει στον νομοθέτη ε, στα πλαίσια νομοθετικών συμφωνιών να πει στους παράγοντε τη αγοράς ότι μια νομοθεσία δεν θα εφαρμοστεί προσωρινά ή λόγω μιας δυσκολίας, ερμηνείας, προσαρμογής κτλ. Νομίζω ότι η λογω μιας δυσκολιας ερμηνεια προσαρμογη κτλ Ένωση δεν χρειάζεται μια τέτοια διαδικασία, γιατί απεδείχθη πολλές φορές ότι μπορούσε να προσαρμόσει την ε, νομοθετική διαδικασία σε πρώτο βάθμιο επίπεδο, δεύτερο βάθμιο επίπεδο και να, προσαρμόσει, να λάβει υπόψη τις ε, συγκυρίες. Και βλέπω αντίθετα μία ανοιχτή πόρτα για όλους τους λομπίστες, για όλους ε, τους παράγοντες των χρηματαγορών που θα βρουν την κερκόπορτα στην νομοθεσία, ούτω ώστε να αναστείλουν την εφαρμογή της. Νομίζω λοιπόν ότι με αυτόν τον τρόπο ε, βάζουμε ήδη μια ρογμή στο μηχανισμό μας, το οπλοστάσιό μας και δεν θέλω κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η θέση μου σήμερα. Θα δούμε όμως σε τι συμβαστική λύση θα καταλήξουμε. Θα ήθελα όμως επευκαιρία να αναφερθώ σε αυτό το πρόβλημα. Επίσης θα πρέπει να βρω μια καλή ισορροπία σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του συστημικού ρίσκου, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Ρίσκου, λαμβάνοντα υπόψη ε, την άποψη τη ε, Συνταγματική Επιτροπή ε, και τη Επιτροπή Προπολογισμών, όπου βασικά θα συζητήσουμε τι, τη διακυβέρνηση. Αν θα πρέπει να τη διευρύνουμε, αν θα πρέπει να περιορίσουμε το ρόλο της, του πρόεδρου τη Κεντρική Τράπεζα ή αυτή η Επιτροπή θα πρέπει να έχει πόρου ικανότητα και όλες τις δυνατότητες της ΕΚΤ και να τις λάβουμε να δώσουμε περισσότερες αυτονομίες λόγω, ε, υπάρχουν, λόγω του ότι υπάρχουν περι, περιπτώσεις να υπάρξει σύγκρουση με την νομισματική πολιτική που διέπεται από την ΕΚΤ. Θα δούμε τι θα γίνει. Αυτές είναι οι αρχικές παρατηρήσεις που ήθελα να κάνω και θέλω συμπερασματικά να σας πω κάτι που, με το οποίο συμφωνώ με τους ε, συνεισηγητές, ότι σε αυτή τη φάση δεδομένου του χρονοδιαγράμματος και της φιλοδοξίας μας η μέθοδος εργασίας θα πρέπει να είναι μία τέτοια που να μας επιτρέπει να συμπεριλάβουμε τους εκπροσώπους των άλλων ομάδων και να δουλέψουμε ομαδικά, συνεργατικά ε, στα πλαίσια της διαπραγματευτικής ομάδας, πέρα από την συνενοχή που έχουμε αναγκαστικά εμείς οι συνεισηγητές. Ευχαριστώ. Thank you. Και εμείς ευχαριστούμε. Από την ομάδα Άλντε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο συνεισηγητές για την εξαιρετική δουλειά που έχουν κάνει μέχρι τώρα. Από την αρχή θα ήθελα να πω ότι αυτές τις ε, χίλιες, χίλιες και κάτι τροπολογίες δεν τις έχω μελετήσει ακόμα. Γι' αυτό η θέση μου δεν έχει διαμορφωθεί ακόμα τελείω, ε, παρά μόνο με βάση τα όσα έχω μάθει και έχω δει ο ίδιος. Ε, όμως ε, είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και έχουμε μεγάλη πρόκληση ενώπιόν μας. Ακριβώς γιατί αυτή η, αυτό το θέμα απαιτεί συνεργασία και έχουμε ήδη μια χρηματοπιστωτική κρίση δεκαετή Έχουμε προβλήματα, έχουμε την, ε, τον αγώνα που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της ενομοποίησης ε, εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ο στόχος πάνω απ' όλα θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον στην Επιτροπή μας ε, να έχουμε ολοκληρώσει τις εργασίες μας μέχρι το τέλος του έτους. Αυτοί οι τρεις τομείς στους οποίους αναφέρθηκε ο συνάδελφος, η αρμοδιότητα, αυτές ε, της ε, Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής, η διακυβέρνηση και η χρηματοδότηση και η Επιτροπή Συστημικού ε, Ρίσκου είναι σωστά χωρισμένες. Για μένα ο συντονισμός πρέπει να γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν πρέπει να προσπαθούμε όπως φοβούνται να δημιουργήσουμε μία εποπτική αρχή παντοδύναμη, αλλά ε, συντονισμό, συντονιστική αρχή. Χρειάζεται λοιπόν ε, η συνεργασία και των εθνικών αρχών, η σύγκριση των ε, εθνικών αποπτικών αρχών, έτσι ώστε να αντλήσουμε διδάγματα και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα και προφανές ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση στην προστασία των καταναλωτών πάνω απ' όλα. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, το σημαντικότερο ίσως. Κάτι το οποίο θα πρέπει ε, να δώσουμε στους ε, πολίτες. Να καταβάλουμε λοιπόν προσπάθειες έτσι ώστε να ενισχυθεί, έτσι ώστε για παράδειγμα ε, να αποσύρουμε από την αγορά επικίνδυνα ε, χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Γι' αυτό θέλει προσοχή και συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αντίθετα τώρα με την Περβάνς ε, δεν ε, συμφωνώ. γιατί, για παράδειγμα, Γνωρίζετε ότι το, στο τέλος του 2019 θα λήξει το Usage Kit. Όμως το PRIPS ε, έχει πολλά προβλήματα ακόμα. Και δεν έχουμε καταλήξει σε μια εκδοχή του με την οποία να συμφωνούμε όλοι. Γι' αυτό λοιπόν ίσως θα έπρεπε να σκεφτούμε να παρατείνουμε την ε, διάρκεια του ΟΣΕΚΑΚΙΤ. Και να μην υποκύπτουμε στις πιέσεις ε, από τα διάφορα λόμπι. Τώρα, μου φαίνεται πως η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή, ιδιαίτερα σε σχέση με τα τρίτα κράτη, θα πρέπει να αναλάβει συντονιστικό ρόλο. Ιδιαίτερα στο θέμα λοιπόν των ισοδυναμιών. Χρειάζεται ενίσχυση της υποχρέωσης κοινοποίησης και διασφάλιση της κάλυψης των κενών ε, στην νομοθεσία στα επίπεδα 2 και 3 τα οποία έχουμε δει στο παρελθόν πως ε, ήταν προβληματικά. Χρειάζεται λοιπόν τροποποίηση και αλλαγή τους έτσι ώστε αυτό, αυτό, αυτά τα κενά να καλυφθούν και τα προβλήματα να διορθωθούν. Τώρα, φοβάμαι πως ε, ανήκω σε μειονότητα για τις ε, απόψεις μου, διότι είμαι υπέρ μιας ε, εκτελεστικής επιτροπής η οποία θα έχει πραγματική εξουσία λήψης αποφάσεων. Αυτό ίσως οφείλεται στη, στον πρώτο επαγγελματικό μου βίο πριν εισέλθω στην πολιτική. Χρειάζεται, κατά την άποψή μου, μια επιτροπή η οποία να μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις και να τις εκτελεί ε, γρήγορα. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να ενισχυθεί και ο ρόλος των καταναλωτών σε αυτές τις επιτροπές. Γνωρίζω πως ε, έχουν ασκηθεί ε, πιέσεις από τα λόμπι για αυτό το θέμα, αλλά θα μπορούσαμε να κοιτάξουμε τις ε, διάφορες λύσεις, να κοιτάξουμε να προβλέψουμε διάφορες αποζημιώσεις. Έχει προταθεί να συνεδριάζει η Επιτροπή αυτή τουλάχιστον πέντε φορές το χρόνο. Για μένα αυτό είναι πολύ λίγο. Θα έπρεπε να συνεδριάζουν τουλάχιστον δύο φορές το μήνα ή και ad hoc όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Σε ό,τι αφορά τώρα τον προπολογισμό έχω υποβάλει τις προτάσεις μου, όμως ε, και πάλι έχω διάφο... Διαφο... Παρακαλώ, έχετε τέσσερα λεπτά, ε, καταλήξτε στα συμπεράσματά σας. Εκτός μικροφώνου, κύριος Κλίντς. Ε, προϋπολογισμός αν θα είναι 35-65% εντάξει αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε. Ποσοστό συμμετοχή τη βιομηχανία του ιδιωτικού τομέα επίσης. Τώρα, ο πρόεδρος ίσως θα χαρεί με αυτό που θα πω. Προτείνω ο πρόεδρος Επιτροπής ΕΚΟ να έχει δικαίωμα ψήφου σε αυτήν την Επιτροπή έτσι ώστε η φωνή του Κοινοβουλίου να εκπροσωπείται. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε για τους πράσινους Φεν Σας ευχαριστώ, προσωπώντας μάλλον τον κύριο Κίχολτ Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συζητητές για το έργο τους. Όσον αφορά τη διακυβέρνηση για τους πράσινους και γενικότερα μιλώντας για την... Έχουμε ως γενικότερη προτεραιότητα να υπάρχει ανεξαρτησία αυτών των τριών αρχών. Θα πρέπει να ενισχυθεί λοιπόν η διακυβέρνηση και των τριών επιγόντως Υποστηρίζουμε λοιπόν την πρόταξη της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου διοικητικού συμβουλίου. Μπορούμε να ε, υποστηρίξουμε τις περισσότερες από οι οποίες έχουν υποβληθεί σχετικά, όμως ο 155 προτείνει να υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης, ενώ η 793 ε, ακόμα και η δυνατότητα πάυσης. Εμείς θα θέλαμε να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο απλό με το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει τη δυνατότητα να, να κοιτάει τους υποψηφίους, υποψηφίους όπως αυτό προβλέπεται στην 736. Με αυτόν τον τρόπο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπει στο ίδιο επίπεδο με, τους, ε, με τον συνομοθέτη, χωρίς να περιπλέκεται η νομοθετική διαδικασία όσον αφορά την προστασία του καταναλωτή και τη διακυβέρνηση. Και εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να ενισχυθεί η εντολή αυτών των οργάνων και να τους δοθούν περισσότεροι πόροι. Κάτι επίσης ουσιαστικό θα ήταν η αντιπροσώπευση των ενδιαφερομένων, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι επαρκής και δεν αμείβεται παρκώς. Αυτό φαίνεται στην έκθεση, στην προσχέδιο της έκθεσης και στις ε, τροπολογίες 663 και 665, 67 ε, και 65. 65. Όσον αφορά τώρα την βιωσιμότητα για το πώς αυτή θα πρέπει να ενταχθεί στο... Θεωρούμε ότι θα πρέπει να ενταχθεί μάλλον στην εντολή της ΕΣΜΑ. Επίσης η ΕΣΜΑ θα πρέπει να αναλάβει περισσότερη δράση για την καταπολέμηση του ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Όσον αφορά την υποπτία τρίτων κρατών, υποστηρίζουμε τις προσπάθειες της ΜΠΕΡΕΣ για την ε, υποπτία των προϊόντων και των υπηρεσιών οι οποίες παρέχονται στην ευρωπαϊκή αγορά από τρίτες χώρες και πιθανώ να δημιουργούν βλάβη. Θα χρειαστεί να έχουμε μια αναρμονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση έναντι των τρίτων χωρών, ιδίω καθώ έρχεται το Brexit, και υποστηρίζουμε τι σχετικέ τροπολογίε που προσπαθούν να το πετύχουν αυτό. Τέλο. Γιατί εγώ SRP για το συστημικό ρίσκο. έχουμε προτείνει να είναι ανεξάρτητο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και υπάρχουν σχετικές τροπολογίες, για παράδειγμα, ε, που αναφέρονται στον διοικητή και στο διοικητικό συμβουλίο της ESRB. Όμω θεωρούμε ότι γενικότερα το ζήτημα του συστημικού ρίσκου θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί στο μέλλον πιο αποτελεσματικά εάν είναι ανεξάρτητη η ESRB. Η SRB έχει υποφεληθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσο καιρό δημιουργεί το. Όμω, αν συνεχιστεί αυτή η σχέση, θα υπάρξουν συγκρούσει συμφερόντων που στην πραγματικότητα αδυνατίζουν την δυνατότητα του ESRB να εφαρμόσει την πολιτική για την προστασία τη φερονγκαιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα συνεισφέρουμε με τι τροπολογίε μα προ αυτήν την κατεύθυνση. που σα είπα, ευχαριστώ του δύο συνεισηγητέ. Ευχαριστούμε. Υπάρχει εκπρόσωπο τη ΓΚΟΕ. FTD. Όχι, η κυρία Κάπελ από το ΕΝΕΦ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους ε, συνεισηγητές. Είναι όντως περίπλοκο το θέμα, αλλά και τεράστια σημασίας. Είναι πολύ λοιπόν ε, σημαντικό, συμμερίζομαι αυτή την άποψη, πώς ε, χρειαζόμαστε επιγόντως μία αναθεώρηση διότι αυτή η έλλειψη συντονισμού και σύγκλησης ε, στην εποπτεία ανάμεσα στα κράτη-μέλη έχει συνεισφέρει ε, στην ε, κρίση σε αυτές τις διαστάσεις που έλαβε. Είναι επομένως σημαντικό η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή να βελτιωθεί. Όπως είπε και ο Ότμαρ Κάρας, χρειάζεται να ενισχύσουμε τη σύγκληση. Επίσης, καλωσορίζω την διαγραφή της άμεσης εποπτείας της ΕΣΜΑ, όπως προβλέπετε στην έκθεση αυτή. Έχει αναφερθεί ότι στην εκτίμηση αντικτήμου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν έχουν, δεν έχουν δημιουργηθεί συμπεράσματα από τα οποία μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το επόμενο βήμα. Ε, πρέπει να φροντίσουμε να μην επιβαρυνθεί η βιομηχανία με υπερβολικά πολύπλοκη νομοθεσία και σε αυτό συμφωνώ με το σχέδιο έκθεσης. Ε, συμφωνώ επίσης και με τις αρμοδιότητες που αναφέρονται ε, με τη διαγραφή της εκ των προτέρων γνωμοδότησης της Επιτροπής. Βέβαια, η πρόταση έτσι όπως ε, αναφέρεται για την υποχρέωση κοινοποίησης και ενημέρωσης ε, στις περιπτώσεις ε, συνεργασίας με τρίτες χώρες με βρίσκει σύμφωνη. Συμμόρφωση, επίσης πολύ σημαντική με, τη, με τα, τις τρίτες χώρες. έχουν συγκεκριμένες διατάξεις, αναφέρονται πολύ συγκεκριμένα λοιπόν στις λεπτομέρειες, γι' αυτό λοιπόν νομίζω πως ε, είναι βάση για να εργαστούμε περαιτέρω. Επίσης η ΕΣΜΑ έχει πολύ σημαντικό ρόλο. Βέβαια, η λειτουργία της θα μπορούσε να γίνεται πιο άμεσα, οι αρμοδιότητες της θα μπορούσαν να είναι πιο άμεσες. Όμως ε, είμαστε υπέρ ε, της ε, ενίσχυσης του ρόλου των εθνικών εποπτικών αρχών. Είμαστε επίσης και υπέρ μιας ανοιχτής διαδικασίας διαβούλευσης όπου χρειάζεται ιδιαίτερα να δοθούν διευκρινήσεις. Τώρα, άρθρο 116β, ε, παράγραφος 2 και 3. Εδώ προτείνουμε να συσταθεί μια τεχνική επιτροπή η οποία θα ε, εργάζεται χωριστά από την ε, πολιτική επιτροπή, διότι το θέμα αυτό αφορά τις τράπεζες και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ τους εισηγητές και όλους τους σκιώδεις εισηγητές. Um, Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα στο Catch the Eye. Κύριε Γκίλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Να σας πω πως έχω αρκετές επιφυλάξεις για τις προτάσεις των εισηγητών και θα ήθελα ορισμένες διευκρινήσεις για κάποιους όρου που προτείνονται για την οκταετή θητεία του Προέδρου της ε, Εποπτικής Αρχής. Υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι υποψήφοι, οι οποίοι δεν επιθυμούν ενδεχομένως να δεσμευτούν για ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Ίσως μια τετραετή θητεία ανανεώσιμη ε, θα ήταν καλύτερη λύση. Έπειτα, παρά το γεγονός ότι προσπαθήσαμε να δούμε ε, τι μπορούμε να κάνουμε στο άρθρο 31α με την, ε, με την ΕΤΑ και τις Εθνικές Εποπτικές Αρχές. Γνωρίζω πως ε, έχουν γίνει προσπάθειες, ε, όμως ε, έχω ακόμα πολλά ερωτηματικά. Υπάρχει σύγχυση. Θα ήθελα λοιπόν ορισμένες διευκρινήσεις σχετικά με το πώς θα προχωρήσουμε. Τέλος, στηρίζω την πρόταση της Περβάνς. Το ξέπλυμα χρήματος θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται στην πρόταση. Στην Επιτροπή Τάξ, μάλιστα, Είχαμε μια συνεδρίαση αφιερωμένη σε αυτό και είναι πολύ βασικό η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή να έχει κάποιες αρμοδιότητες στο τομέα αυτό, στο ξέπλυμα χρήματος. Ευχαριστώ. Θα ήθελα κάποιος άλλος το λόγο. Οι συγκητέ, ο λόγος εσά. Ποιος θα ήθελε να αρχίσει. Α, θέλετε το λόγο. Τον έχετε. Thank you, Chair. Sorry for being late. Ευχαριστώ που καθυστέρησα. Ήμουν στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ, ευχαριστώ τους συναδέλφους για τον εντυπωσιακό όγκο τροπολογιών που υποβλήθηκαν. Θέλω να σταθώ σε κάποιες που αφορούν τις σχέσεις ε, με τη διεύθυνση. Καταρχάς, ε, για τις αναφορές. Μετά την ολοκλήρωση του κειμένου, ε, είδαμε ότι δεν υπάρχει αρκετή σαφήνεια για τα ε, ρυθμιζόμενα ε, στοιχεία αναφοράς των και για να το ε, λύσουμε, προτείναμε τρει τροπολογίε για να εξασφαλίσουμε ότι τα, τα, οι όροι αναφορά ή τα κινητά data μπορούν να χρησιμοποιούνται στην Ένωση και ότι δεν θα υπάρχει διαταραχή στην αγορά χωρίς να ε, υποσκάπτουμε τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την ε, διακυβέρνηση στα benchmark. Επίσης, τα critical benchmark, όπως και το Euribor. Έχω δουλέψει στη σχετική ομάδα, ε, ούτως ώστε να υπάρξει μια ομαλή μετάβωση σε πιο αξιόπιστη κατάσταση. Ε, όμως, για τα critical benchmark χρειαζόμαστε ε, μια μεγαλύτερη μεταβατική περίοδο για να υπάρχει ομαλή μετάβαση. Μια επέκταση κατά δύο χρόνια της μεταβατικής περίοδου θα επιτρέπει ε, ελάχιστη διαταραχή της αγοράς και θα μειώσει το κίνδυνο για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Επομένως, θα ήθελα να καλέσω όλους σας να συμπεριλάβετε τις τροπολογίες, του συμβασμού και να οριστικοποιήσετε τουλάχιστον ω τμήμα της α, αναθεώρησης των Ευρωπαϊκών Αποπτικών Αρχών το συντομότερο δυνατόν ε, να τα βάλετε αυτά τα στοιχεία λοιπόν. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν θέλει να πάρει το λόγο. Thank you very much, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ όλους σας στο Κοινοβούλιο για την υποστήριξή σας. Ε, τη χρειαζόμαστε για αυτό το φάκελο και ευχαριστώ για τις προτάσεις που μας κάνατε. Ακόμα εξετάζουμε τις τροπολογίες. Από την σημερινή συζήτηση θα ήθελα να σταθώ σε τρία θέματα τα οποία έθεσαν διάφοροι. Καταρχά Καταρχάς είναι για το, την καταπολέμηση του ξαπλήματος του χρήματος. Ε, πριν από λίγες εβδομάδες κάναμε αυτή την πρόταση. Ε, θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό, κάτι πρέπει να γίνει και διαβάζουμε στον τύπο ότι υπάρχουν όλο και περισσότερα στοιχεία, ότι πρέπει να γίνει κάτι γρήγορα στον τομέα αυτό της καταπολέμησης του ξεπλήματος. Έχει απόλυτο νόημα να γίνει μαζί με την αναθεώρηση των Ευρωπαϊκών Υποπτικών Αρχών Γι' αυτό παρουσιάσαμε την πρόταση ω τροπολογία στην πρόταση για την αναθεώρηση των αρμοδιοτήτων των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών. Είναι αλλαγέ οι οποίε γίνονται πέρα ε, και επιπλέον από την αναθεώρηση των ΕΖΑ, των Ευρωπαϊκών Υποπτικών Αρχών, για τη διακυβέρνηση και για τις αρμοδιότητες που έχουν όλες αυτές οι υποπτικές αρχές. Πιστεύουμε λοιπόν ότι τα δύο στοιχεία ε, πρέπει να πάνε παράλληλα. Δεύτερον, για την προστασία των καταναλωτών θεωρώ ότι είναι ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό εδώ στο Κοινοβούλιο και συμφωνούμε κι εμείς. Έγιναν προτάσεις για τις ε, αρμοδιότητες ε, για την παρέμβαση προϊόντων και είναι σημαντικό να ενισχύσουμε την ε, σημασία των μέτρων αυτών για την παρέμβαση που έχει έσμα σε προϊόντα και πώς θα ενισχύσουμε αυτές τις αρμοδιότητες. Και το τρίτο είναι ε, για το No Action Letter. Ε, καμία δράση από την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς, δηλαδή. Είναι μια ιδέα η οποία ακούστηκε πιο πρόσφατα στη συζήτηση ε, και δεν είναι εύκολο να εφαρμοστεί νομικός πώς. Ε, είχαμε συζητήσεις με, τους, με την νομική υπηρεσία και σας λέω από τώρα ότι δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει ε, με οριζόντιο τρόπο στους ε, ιδρυτικούς κανονισμούς. Υπάρχουν κάποια εργαλεία που έχουν οι εποπτικές αρχές στην τομεακή νομοθεσία και οι εποπτικές αυτές αρχές έχουν την εξουσία, την αρμοδιότητα να ξεκινήσουν μια αναθεώρηση ενός μέτρου επίπεδου 2 εάν δουν ότι υπάρχει μια εξέλιξη στην αγορά που το καθιστά αναγκαίο. Το να το έχουμε όμως ως οριζόντιο μέτρο ε, στον ιδρυτικό κανονισμό ε, είναι δύσκολο να εφαρμοστεί νομικός πώς. Ευχαριστώ πολύ. Πριν δώσω τον λόγο στους εισηγητές θα Ε, να πω κι εγώ. Αυτό που είπε για την τροπολογία του Προέδρου της, ε, ε για τον Πρόεδρο της Επιτροπής ΕΚΟΝ ως τμήμα της Διευθύνουσας Ομάδας, ε, δεν έχω επίσημη θέση, αλλά έχω ε, κάποιες αμφιβολίες για το κατά πόσον ο νομοθέτης πρέπει να είναι και μέλος ενός συμβουλίου, ας πούμε, σε αυτές τις αρχές, τις υποπτικές αρχές. Ε, για την πρόταση του κ. Μπάλτ και των Πρασίνων για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, όπου σας καλώ να είμαστε προσεκτικοί για να μην αλλάξουμε την ισορροπία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο φορέα αυτό που τον υποστηρίζει η Εγώ προτείνω ε, ο επικεφαλής της γραμματείας να αναβαθμιστεί ο, ο ρόλος τους, να ψηφίζει στη διευθύνουσα ομάδα και στο Γενικό Συμβούλιο, βεβαίω, ναι, το δέχομαι, αλλά αν βάλουμε μια διαδικασία όπως αυτή του διευθυντή, ας πούμε, αλλάζει η ισορροπία. Και θα πρέπει να σκεφτούμε την περίπτωση ε, το Συμβούλιο αυτό να μην εδράζεται στο εσωτερικό της ΕΚΤ. Να μην, να μην ανήκει στην ΕΚΤ πια. Δεν θέλω να ε, επιβάλλω έναν ακόμα θεσμικό μια θεσμική περιπλοκή σε αυτό το περίπλοκο θεσμικό πλαίσιο. Σκεφτείτε το. Εσείς οι συγητές και ας το σκεφτεί και η διαπραγματευτική ομάδα και τώρα οι συνεισηγητές μας για τις καταληκτικέ παρατηρήσεις υπερβάνς ε, Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και εσάς και τους υπόλοιπους συναδέλφους που τοποθετήθηκαν. Πρέπει να εξετάσουμε κάθε ανησυχία, κάθε σχόλιο έτσι ώστε να συνεργαστούμε παρά το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, όταν υπάρχουν καλές προθέσεις, ε, νομίζω πως ε, αυτό βοηθά. Πρέπει να σκεφτούμε ποιες είναι οι συνέπειες αυτών που φανταζόμαστε εμείς εδώ, αυτόν που προσπαθούμε να κάνουμε. Πρέπει να αναλογιστούμε τις επιπτώσεις και τις διασυνδέσεις ανάμεσα ε, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, σε, στις ευρωπαϊκές αρχές και στο Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου. Γι' αυτό λοιπόν ε, σας ευχαριστώ για όλες τις προτάσεις. Τώρα για την ε, θητεία την οκταετή. Η εμπειρία μου έχει δείξει πως η ανεξαρτησία της ε, αρχής είναι ε, μεγαλύτερη στη δεύτερη περίοδο ε, θητεία, στη δεύτερη θητεία παρά στην πρώτη. Όταν δηλαδή ξαναδιορίζονται είναι καλύτερα τα πράγματα. Η ανεξαρτησία λοιπόν πρέπει να διασφαλίζεται πάση θυσία. Το έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει ε, και νομίζω πως πρέπει να σταθούμε εκεί. Ε, ε, τόσο ως προς τον έλεγχο, όσο και ως προς την ίδια την ανεξαρτησία τώρα. Η Επιτροπή που θα ασχολείται με το ξέπλυμα χρήματος. Υπάρχει ήδη Επιτροπή με αυτές τις αρμοδιότητες. Σας ευχαριστούμε πάντως πάρα πολύ για όλες τις προτάσεις σας. Τις έχουμε λάβει όλες. Τώρα, τέλος αυτής της εβδομάδας, αρχή της επόμενης, οι συντονιστές θα πιάσουν δουλειά. Θα συνεργαστούμε και με τις ε, άλλες συνδεδεμένες επιτροπές. Θα ζητήσουμε γνωμοδοτήσεις και από την Επιτροπή Λίμπε, για παράδειγμα. Φυσικά πρέπει να γίνει διάλογος Και φυσικά υπάρχουν ε, διαφορές, υπάρχουν δύο ξεχωριστές εκθέσεις, όμως ε, συνδέονται μεταξύ τους. Γι' αυτό θεωρώ πως πρέπει να δούμε το όλο θέμα ως ένα σύνολο και να μην χωρίσουμε και κατακαιρματίσουμε την έκθεση αυτή. Να μην γίνονται παράλληλες συζητήσεις, έτσι ώστε να ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας και για τους δύο φακέλους το συντομότερο. Και η συνεισηγήτριά μου και εγώ θα χρησιμοποιήσουμε όλο το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Την Πέμπτη θα συναντηθούμε, οι σκιώδες εισηγητές, έτσι ώστε να ε, διοργανώσουμε συνάντηση σκιωδών μέσα στον Οκτώβριο. Σας ευχαριστώ πολύ. και στις τροπολογίες, τις οποίες ε, σχεδόν όλες έχω διαβάσει, έτσι, αλλά και στις ε, προφορικές παρεμβάσεις, υπάρχουν σημεία δυσκολίας. Επιβεβαιώνονται αυτές τις δυσκολίες, λοιπόν. Υπάρχουν όμως και διάφορες ιδέες, ε, διάφορες τάσεις που προκύπτουν, που μας επιτρέπουν να βελτιώσουμε την πρόταση της Κομισιόν και να φτάσουμε σε καλό κείμενο. Υπάρχει ένα σημείο το οποίο δεν ακούστηκε, δεν αναφέρθηκε και όμως είναι σημαντικό. Είναι η συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, στην, και με την πρωτοβουλία των συνεισηγητών, αλλά και με τις συνεισφορές των διαφόρων ευρωβουλευτών σε όλο το σύστημα των κατευθυντήριων γραμμών, των συστάσεων, των ερωταποκρίσεων, επί των οποίων δεν έκανε πρόταση η Κομισιόν, αλλά λόγω της πλούσιας εμπειρίας του, το Κοινοβούλιο μπορεί να συνεισφέρει με αυτούς τους τρόπους. Διάφορες ε, παρεμβάσεις στάθηκαν στο ρόλο των ισοδυναμιών, στην κατάσταση δηλαδή που υπάρχει στις τρίτες χώρες. Με τον κύριο Μπάλς βάλαμε επιτάπητος ένα βασικό σημείο ισορροπίας μεταξύ των συνεισηγητών για το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα της ισοδυναμίας. Κατά τα άλλα, η πρόταση της Κομισιόν, η οποία συνδέει στενά τις αρχές αυτές με την ε, αξιολόγηση για τη χορήγηση της ισοδυναμίας, αυτό είναι, λέει η Κομισιόν εκ των Όνου και αυτό το ρόλο το ενισχύουν κάποιες τροπολογίες έτσι στο θέμα της α, εκχώρησης αρμοδιοτήτων. Η πρόταση τη Κομισιόν είναι υπερβολική. Αλλά νομίζω ότι η ιδέα ότι πρέπει να υπάρχει μια κοινοποίηση και μια δυνατότητα να εντοπίζουμε την γεωγραφική προέλευση, συγγνώμη, για τις αντιπροσωπείες μάλλον, από πού προέρχονται γεωγραφικά, νομίζω γίνεται. Ε, για την προστασία των καταναλωτών έχουμε πολλές α, ε, τροπολογίες. Και εγώ έχω υποβάλει σχετικέ τροπολογίε, ούτω ώστε να έχουμε περισσότερε δυνατότητε ε, αναστολή ή απαγόρευση προϊόντων τα οποία είναι επικίνδυνα για του καταναλωτέ. Αυτή είναι μια καλή βάση. Και για την ιστορία των 8 χρόνων, τη 8 ε, συμφωνώ με τον προλαλήσαντα. Και μάλιστα να προσθέσω ότι θεσμικός πώς και από τη σκοπιά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν υπάρχει μια ανανέωση της θητεία, βλέπουμε ότι η τάση είναι να μην βλέπουμε, ας πούμε, να μην ψάχνουμε νέες αρμοδιότητες και ε, πραγματογνωμοσύνη, αλλά ουσιαστικά να βασιζόμαστε ε, στα παλιά, ας πούμε, να κάθομαστε στα αυγά μας. Ε, επομένως, σε αυτή την περίπτωση ε, θα πρέπει να παίξει βασικό ρόλο το Κοινοβούλιο ε, στην ανανέωση της θητείας δηλαδή. Τώρα, για τα διάφορα προϊόντα δεν, προ... δεν ε, μίλησα στην αρχική μου παρέμβαση. Επιβεβαιώνω τη θέση που λάβαμε με τον κύριο Μπάλς. Προτείναμε δηλαδή την απόσυρση διαφόρων προϊόντων και την άμεση εποπτεία, αντίθετα από ό,τι έκανε η Κομισιόν. Για το ανημερωτικό φυλάδιο θα πρέπει να δούμε τι είναι δυνατόν να κάνουμε και τι όχι, γιατί υπάρχει μια βάση η οποία μπορεί να είναι χρήσιμη εδώ και σημειώνω ότι για τις, τους όρους αναφορά στα benchmark υπάρχουν διάφορες τροπολογίες που κατατέθηκαν. Δεν είμαι σίγουρη ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την πρόταση για να ξανανοίξουμε την νομοθεσία για τα benchmark ε, αυτή καθεαυτή. Αλλά σε αυτό που προτείνει η Κομισιόν θα πρέπει να προσαρμόσουμε τις προϋποθέσεις εποπτείας. Αυτά. Χαίρομαι που θα συνεργαστούμε, θα δουλέψουμε μαζί και ελπίζω να μπορέσουμε να ψηφίσουμε στην, Ευρωπαϊκή, Επιτροπή μας ε, πριν το τέλο του 2018, ούτω ώστε να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, που ελπίζω επιτέλους να ανασκουμποθεί και να επιταχύνει τι εργασίες του. Σα Σας ευχαριστούμε. Συμφων... Ε, έχω και εγώ την ίδια ελπίδα με εσά. Να σας ενημερώσω ότι 5 Νοεμβρίου έχει... είχε προγραμματιστεί και συνεχίζει να είναι αυτός ο προγραμματισμός, αν και είναι υπερβολικά αισιόδοξο για την ψηφοφορία στην ΕΚΟΝ. Βεβαίω θα μας ενημερώσει η συγγετρία σχετικά. Γνωρίζουμε ότι η Επιτροπή προσπαθεί να επιταχύνει τη διαδικασία έτσι ώστε να γίνουν ουσιαστικοί τριμερείς διάλογοι και ενθαρρύνουμε και το Συμβούλιο να δείξει και αυτό την ίδια αποφασιστικότητα με αυτή που φάνηκε στη σημερινή μα συνεδρίαση και συζήτηση. Σα ευχαριστώ. Α περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξη. Είναι η ετήσια έκθεση για τι οικονομικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η συγγήτρια Μπάρμπαρα Κάπελ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξαιτία της ε, πολυμορφίες των δραστηριοτήτων τη Ευρωπαϊκή Τράπεζας Επενδύσεων και του μεγάλου χαρτοφυλακίου της, ε, το έργο που έχουμε αναλάβει είναι πάρα πολύ φιλόδοξο. Το πρώτο σχέδιο είναι σε αρχικό στάδιο κόμμα. Θα με χαρώ πολύ να λάβω τις ε, τροπολογίες σας ε, και θα ήθελα να πω ότι χρειαζόμαστε ένα καλύτερο σχέδιο. Θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω τους, ε, το ΕΛΚΑ όχι μόνο γιατί φρόντισε να πάρουμε στοιχεία και από, και από το Λουξεμβούργο, αλλά ε, και επειδή φρόντισε να είναι εδώ πρόσωποι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και ίσως ε, αυτό να μας δώσει τη δυνατότητα να ακούσουμε και την άποψή τους. Το σχέδιο έκθεσης χωρίζεται σε 8 κεφάλαια. Αναφέρεται στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής ε, Τραπέζας Επενδύσεων. Φέτος είναι η επέτειος 60 ετών ε, της ΕΤΕΠ και στο σχέδιο έκθεσης αναφέρει ορισμένα από τα επιτεύγματα της ΕΤΕΠ αυτά τα 60 χρόνια λειτουργίας της. Έχουν γίνει επενδύσεις μέχρι τώρα 11, σε 11.800 11, project σε πολλές χώρες αξίας 1.100 ε, ε, δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι εντυπωσιακά τα ποσά αυτά, εντυπωσιακή και η επίδοση του ΕΦΣΥ, το οποίο Έχει εγκρίνει 898 project αξίας 335 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό λοιπόν έχει οδηγήσει και στην ε, παράταση του ΕΦΣΙ, στο ΕΦΣΙ 2 δηλαδή, μέχρι το 2020. Ε, παρά τις αμφιβολίες ε, ορισμένων στην αρχή της ε, πορείας του. Νομίζω πως το ΕΦΣΙ είναι ένα επιτυχημένο project. Επίσης, αναφέρομαι στην ε, διαφοροποίηση των επενδύσεων, σε, στην καινοτομία, στο περιβάλλον, υποδομές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηρίζονται ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την ΕΤΕΠ διότι η στήριξη αυτή είναι απολύτω σημαντική για την ίδια την ύπαρξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επίση, είναι πολύ σημαντικό ε, να, ε, έχει, να υπάρχει ειδικό κεφάλαιο αφιερωμένο στην ε, Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ανθεκτικότητας, ERI, να γίνεται ιδιαίτερη μνήμα στην μεταναστευτική και προσφυγική κρίση και στην καταπολέμηση των αιτίων της. Έχουν εγκριθεί μέχρι τώρα 26 ε, project από την ERI αξίας 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σύνολο δημιουργία 100.000 100.000 ε, θέσεων εργασίας μέσω των ε, χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΡΙ. Ε, είναι πολύ σημαντικό και για την δημιουργία θέσεων απασχόλησης και για τη δημιουργία υποδομών στις χώρες ε, διέλευσης και για ε, τους ίδιους τους ε, μετανάστες και τη στήριξή τους. Επίσης υπάρχει ξεχωριστό κεφάλαιο για το Brexit. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ποσοστό 16,1% συμμετοχής στο ταμείο αυτό. Χρειάζεται λοιπόν ε, μια συμφωνία ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο για την ε, αποπληρωμή αυτού του ποσού. Αυτή τη στιγμή είναι επίσης σημαντικό να δούμε τι θα γίνει και με τους ε, υπαλλήλους, με τους συνεργάτες μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Φέτος το Σεπτέμβριο εκδόθηκε ένα ομόλογο 500 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της ευγεσιμότητας και των ε, στόχων. Μιλώσαμε ένα, ένα ομόλογο για την πράσινη ανάπτυξη. Το δεύτερο σημείο που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό είναι η χορήγηση πιστώσεων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΤΕ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο εδώ το 2017 χρηματοδοτήθηκαν 100 νέα project ε, με ποσό αξίας 7,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι τρίτες χώρες έλαβαν στήριξη 23 δισεκατομμυρίων ευρώ. Επίσης, ε, το SCP Investment Facility ε, είναι σημαντικό να αναφερθεί η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αφρική που χρηματοδοτείται από την ΕΤΕΠ και ε, η δράση της ΕΤΕΠ για την προστασία των πρώτων υλών στην Αφρική. Επίση, γίνεται αναφορά στη συμμόρφωση τον Ιανουάριο. Η ΕΤΕΠ ανέλαβε την καταπολέμηση της ε, φορολογικής απάτης, φοροαποφυγής, φοροδιαφυγής, επιθετικής φορολογικής πολιτικής. Beneficial ownership είναι και αυτό μέσα στην έκθεση. Αυτά λοιπόν πολύ συνοπτικά από μένα. Θα χαρώ πολύ για την συνεργασία με τους εσκιώδεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριος Λάγκεν για το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ την ε, εισηγήτρια. Μας έδωσε όντως πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και νούμερα για τις ε, τρέχουσες δραστηριότητε της ΕΤΕΠ. Το σχέδιο έκθεσης είναι αρκετά καλό, πολύ καλό θα έλεγα. Το λέω εδώ και καιρό. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει αναφορά και μάλιστα θα μπορούσε να γίνει η έκθεση δύο πρωτοβουλία για την 60η επέτειο της ΕΤΕΠ διότι ε, πρέπει να μην ξεχνάμε ότι εδώ γίνονται πράγματα και εμείς ε, δεν πρέπει να καθόμαστε και να θεωρητικολογούμε. Ορισμένες παρατηρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, αύξησε το κεφαλαιά της τα τελευταία χρόνια είναι το μόνο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα διεθνές στο οποίο συμμετέχουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη με προϋποθέσεις σε διάφορους τομείς. Για παράδειγμα, ελάχιστο ποσοστό 25% επενδύσεων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και για την προστασία του περιβάλλοντος. Η ΕΤΕΠ επίσης Διατραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στις ε, εξωτερικές δραστηριότητες, στην αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το είπε και η κυρία Κάπελ αυτό, ε, μέσω των διαφόρων πρωτοβουλίων που στηρίζει. Και ε, αυτό είναι κάτι που το καλωσορίζουμε και ελπίζουμε να διατηρηθεί σε συνεργασία με τις εθνικές επενδυτικές τράπεζες με την Παγκόσμια Τράπεζα, με την Παγκόσμια Τράπεζα Ανάπτυξη της Ασίας ε, έχουν δείξει πολύ σημαντικό έργο. Γι' αυτό χρειάζεται να στηρίξουμε την ΕΤΕΠ έτσι ώστε να διατηρήσει την, ε, τις ισορροπίες, να μην ανταγωνίζεται τις ε, εμπορικές τράπεζες, αλλά αντίθετα να φροντίζει για ίσους όρους ανταγωνισμού. Επίσης, όπως είπε και η κυρία Κάπελ, είναι πολύ, σημαντικό, πολύ σημαντική αναφορά στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής, των ε, υψηλών ε, προτύπων ε, της ΕΤΕΠ. Γνωρίζουμε ότι ορισμένα project είναι πολύ σημαντικά και ασκείται μεγάλη πίεση στην ΕΤΕΠ για χρηματοδότηση. Σίγουρα πρέπει να θωρακίσουμε την ΕΤΕΠ από αυτέ τι πιέσει, όμως ελπίζω πως με τους άλλους σκιώδει εισηγητέ και με την ε, εισηγήτρια κυρία Κάπελ θα καταλήξουμε σε μια έκθεση καλή, μέλλοντο στραφή και ε, συμπαγή. Σας ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε για την Άλντε. Ε, να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω γιατί οι συνάδελφοι από τους σοσιαλδημοκράτες αποχωρούν από την αίθουσα κάθε φορά που ε, παρουσιάζει η κυρία Κάπελ έκθεση. Ε, αυτό δεν είναι ε, σωστή συμπεριφορά. Υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος των σοσιαλιστών, κάποιος συνάδελφος να Και εσεί, κύριε Πρόεδρε ανήκετε στου σοσιαλδημοκράτε. Βλέπω ότι βγήκαν όλοι έξω και δεν είναι πρώτη φορά που το παρατηρώ αυτό. Είναι μια στρατηγική που κρύβεται από πίσω. Δεν, δεν γίνεται να δουλεύουμε έτσι. Actually, uh, there are more... Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή στην αίθουσα υπάρχουν περισσότεροι συνάδελφοι από του σοσιαλιστέ, παρά από το ΕΛΚ. Θα αναρωτιόταν κανεί γιατί οι συνάδελφοι του ΕΛΚ δεν είναι παρόντες όταν μιλάει ο συνάδελφο του. Ε, κύριε Πρόεδρε, μην μη με περνάτε για βλάκα. Τα βλέπω αυτά με τα μάτια μου. There are three όχι, όχι, δεν σα περνάω για τίποτα. Απλώ τρει συνάδελφοι από του σοσιαλιστέ βρίσκονται στην αίθουσα αυτή τη στιγμή. Ε, λογική ίσω να είναι ερώτησή σα, αλλά όχι αυτή τη στιγμή να μην είναι η καταλληλότερη για να τη θέσετε. Αφήστε το. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, εκπροσωπώ τον συνάδελφο κύριο Κόχλι. Ναι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Κάπελ για την ε, καλή τη έκθεση. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιε. Ε, κάποιοι τομείς στους οποίους μπορεί να βελτιωθεί. Σε αντίθεση με άλλες τράπεζες, το 100% της, ΕΚ, της ΕΤΕΠ βρίσκεται στα χέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε τον πλήρη έλεγχο. Θα θέλαμε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση πολιτικών για την ανάπτυξη. Θα πρέπει επίσης ταυτόχρονα η ΕΤΕΠ να ενισχύσει περισσότερο την βελτίωση των διοικητικών δυνατοτήτων και την ε, αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης των διαφορών κρατών μελών, γιατί αυτή έχει τεράστιο, τεράστια σημασία και για τους πολίτες και για την οικονομία. Η ΕΤΕΠ θα πρέπει επίσης να ενισχύσει περισσότερο τις δραστηριότητες επικοινωνίας, δημοσιοτήτα του έργου της προς το κοινό. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να υπάρξει μεγαλύτερη δυνατότητα παρέμβαση των πολιτών, έτσι ώστε και εκείνοι να έχουν λόγο. Με αυτόν τον τρόπο, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να έρθει πιο κοντά στους πολίτες της. Είναι επίσης σημαντικό να σημειώσουμε ότι έχουμε ένα σύστημα διακυβέρνησης, οικονομική, διακυβέρνησης περίπλοκο, το οποίο θα πρέπει να αξιοποιήσουμε πιο αποδοτικά και με μεγαλύτερη συνεκτικότητα στον τρόπο με τον οποίο επιλέγονται τα project που χρηματοδοτούνται και ποια είναι η σχέση αυτών των project με τις συστάσεις αναχώρα και τις μακροοικονομικές προοπτικές τους. Η ΕΤΕΠ επίσης θα πρέπει να ενισχύσει τη χρηματοδότηση των ε, έργων τα οποία υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο και συνδέονται με την τοπική κοινωνία. Επίσης θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος εποπτείας της ε, ΕΤΕΠ, όχι μόνο από την ΕΚΤ, αλλά χρησιμοποιώντας και εκπροσώπους της ΕΣΜΑ, της ε, πιθανώς εξωτερικούς και της EBA, εκτός από την ΕΚΤ. Σας ευχαριστώ. Thank you. Και σας ευχαριστούμε κύριος Παπαδημούλης. Ε, ε, είστε έτοιμος κύριε Παπαδημούλη να πάρετε το λόγο. Για την ΚΟΕ, λοιπόν, ο κύριος Παδημόλης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη γιατί ήρθα κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, αλλά μόλις τελείωσε το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, ε, αλλά πιστεύω ότι χρειαζόμαστε μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση για την ε, έκθεση που θα πρέπει να ετοιμάσουμε για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ε, και νομίζω ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε και προτάσεις που είχαμε ετοιμάσει και τα προηγούμενα χρόνια ε, για αυτό το θέμα γιατί είμαστε σε μια φάση που χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις γιατί υπάρχουν περιφέρειες και κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου έχει ενταθεί η αποεπένδυση, γιατί υπάρχουν μεγάλα επενδυτικά κενά, γιατί πρέπει να επενδύσουμε πολύ περισσότερο στην καινοτομία, στις επενδύσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον, την κυκλική οικονομία, την πράσινη οικονομία. Και ο ρόλος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων μπορεί να συμβάλλει πολύ και στο στόχο μιας διατηρήσιμης, δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης. Σκοπεύω εκ μέρους πολιτική μου ομάδας να καταθέσω τροπολογίες ε, στην ε, έκθεση που μας ε, παρουσιάστηκε και επίσης να συνεργαστώ όχι μόνο με την εισηγήτρια αλλά και με τους σκιώδεις εισηγητές και των άλλων πολιτικών ομάδων προκειμένου να βελτιώσουμε το κείμενο το αρχικό που μας έχει κατατεθεί. Σας ευχαριστώ. thank you. As there are no other... Σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω να ζητάει ε, το λόγο κάποιος άλλος συνάδελφος. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Μετήσεων, τον κύριο Ντοκέλεβιτς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύντομα, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Κάπελ και όλα τα άλλα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εμπλέκονται σε αυτή τη συζήτηση να σας ενημερώσω ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μεταμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια. Βέβαια δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο και επ' αυτού θα συμφωνήσω με τον κύριο Παπαδημούλη ότι πράγματι χρειάζεται να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για επένδυση στην Ευρώπη αν δούμε τα δεδομένα. Το ποσοστό επένδυσης στην Ευρώπη είναι κατά 10% μειωμένο σε σχέση με το 2007 σε πολλούς τομείς, ιδιαίτερα για παράδειγμα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την ψηφιακή οικονομία, ε, ψηφιακή μετάβαση, είναι τομείς στους οποίους έχουμε σημαντικές προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε. Η ΕΤΕΠ έχει υλοποιήσει ουσιαστικά το πρόγραμμα ΕΦΣΥ και είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό. Έχουμε και πολλές προκλήσεις μπροστά μας. Μία από τις δυσκολότερε είναι το Brexit και θα πρέπει να βρεθεί ένα τρόπο ανα, ε, ανακεφαλαιοποίηση για να καλυφθούν τα κεφάλαια που θα χαθούν από την έξοδο τη Μεγάλη Βρετανία. Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Υπάρχει μια διαδικασία διαβούλευση με του μετόχου. Ε, Όμω αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί γρήγορα και ελπίζω αυτό να γίνει το συντομότερο δυνατό γιατί πρέπει να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τις αγορές ε, που να τους αποδεικνύει ότι το μοντέλο, ε, το επιχειρηματικό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είναι βιώσιμο. Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό να το διασφαλίσουμε μετά το Brexit. Ε, μια άλλη μεγάλη πρόκληση είναι οι διαπραγματεύσεις που γίνονται για το πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Εμείς υποστηρίζουμε την ιδέα ότι η δομές διοίκηση, οι οποίες λειτουργήσαν αποτελεσματικά για το ΕΦΣΥ θα πρέπει να διατηρηθούν. Η κυρία Βέρν... Βέρνικε είχε αναφερθεί στο ρόλο που έχει να παίξει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την Ανάπτυξη. Ε, είμαστε μια ευρωπαϊκή τράπεζα και γι' αυτό οφείλουμε να εφαρμόζουμε την ε, πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, δεν θα έλεγα ότι αυτή την άποψη, αυτή την οτροπία την αντανακλούν όλε οι διάφορε προτάσει οι οποίε έχουν υποβληθεί. Σε συνεργασία λοιπόν με του συνομοθέτε, ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε λύσει ε, για να μην υπονεμευτεί ή να μην αποστοχωρήσουμε σε τίποτα από αυτά που λειτουργούν στην πραγματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πιο συγκεκριμένα ο δανεισμός, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη σημασία και για, τις, για τα κράτη-μέλη και για την ε, ε, Κεντρική Τράπεζα ε, και για όσου υλοποιούν project χρηματοδοτούμενα από την ΕΤΕΠ. Όταν κάποια πράγματα λειτουργούν καλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τα προστατεύουμε. Θα έλεγα ότι εμείς προσπαθούμε να προωθήσουμε σε μεγάλο βαθμό τα έργα τα οποία έχουν τοπικό αντίκτυπο, έχουμε εταιρικέ σχέσεις με τις περιφερειακές αρχές, με εθνικά ε, Ινστιτούτα, ε, τράπεζες ή εργαλεία για την περιφερειακή ανάπτυξη. Έχουμε ε, συγκεκριμένα δάνεια για τα περιφερειακά προγράμματα και διάφορα χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για την εφαρμογή των, σε συνδυασμό με τα διαρθρωτικά ταμεία. Χωρίς να μπω στις λεπτομέρειες, θα έλεγα ότι με τις αλλαγές που έχουν γίνει στο, στον ε, δημοσιονομικό κανονισμό, που και αυτός Αυτέ οι αλλαγέ ολοκληρώθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με αυτέ τι αλλαγέ, λοιπόν, μπορέσαμε να ε, χτίσουμε ε, χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κοινού με τα διαρθρωτικά ταμεία. Κατά τα άλλα, θα συμφωνήσω μαζί σα ότι όσον αφορά τη δημοσιότητα προ τα έξω δεν είμαστε και τόσο αποτελεσματικοί. Δεν ξέρω και πώ μπορεί αυτό να λυθεί. Ε, είναι οδυνερό, αλλά το αναγνωρίζω. Ε, προσπαθούμε πάντω να το διορθώσουμε. Κύριε Πρόεδρε, αυτά από τη μεριά μου και βεβαίω ευχαρίστω να απαντήσω ερωτήματα των Ευρωβουλευτών, αν υπάρχουν. Ευχαριστώ πολύ. Η συγκεκριμένη έχει το λόγο. Κύριε Κάπελ, σα ευχαριστώ πολύ. Βλέπω ότι 6.000 χαρακτήρες δεν φτάνουν για μια τέτοια έκθεση που αφορά την ε, ΕΤΕΠ. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό όλα αυτά που είπαν οι συνάδελφοι, όλη η συμβολή των ε, σχεδόν συγχυτών να ε, συμπεριληφθεί, να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Στο παρελθόν δυστυχώ, δυστυχώς έχουμε κάνει λάθη, πρέπει όμως να φροντίσουμε να συμπεριληφθούν όσο δυνατόν περισσότερες απόψεις σε αυτό το περιορισμένο χώρο των 6.000 χαρακτήρων. Με μεγάλη μου χαρά λοιπόν θα λάβω απόψη τις ανησυχίες σας. Είναι σίγουρα στήριξη της πράσινης οικονομίας, της κυκλικής οικονομίας, ιδιαίτερη έμφαση στην συμμόρφωση, ε, στο beneficial ownership και σίγουρα δεν πρέπει να μείνουμε μόνο στα λόγια, αλλά να περάσουμε στις πράξεις. Ε, επίσης, ε, έχω γνώση του ότι η χρηματοδότηση ε, έργων σε τρίτες χώρες είναι ιδιαίτερα σημαντική, ιδιαίτερα σε αναπτυσσόμενες χώρες οι οποίες ε, χρειάζονται τη στήριξη της ΕΤΕΠ για ε, την επιτυχία των έργων αυτών. Είναι μια τεράστια ευκαιρία όχι μόνο για τις χώρες αυτές αλλά και για την ευρωπαϊκή οικονομία με την έννοια της ε, βιωσιμότητας και της ενίσχυσης της Αφρικανικής Υπήρου, ιδιαίτερα ε, σε σχέση με την στρατηγική της Ένωσης για την Αφρική. Ελπίζω λοιπόν να συνδυάσουμε όλες τις συνσφορές σας, να καταλήξουμε σε μια πλούσια έκθεση η οποία θα σταθεί αντάξια του έργου και της ιστορίας της ΕΤΕΠ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τροπολογίες έχουμε μέχρι τι 11 Οκτωβρίου, θα εξετάσουμε τις τροπολογίες στις 12 Νοεμβρίου, θα ψηφίσουμε στην ΕΚΟΝ 19 Νοεμβρίου. Και προχωρούμε στο επόμενο σημείο. Η Εβάνα Μαλέτιτς έχει ετοιμάσει ένα σχέδιο γνωμοδότηση για τι κοινέ διατάξει. για τα ευρωπαϊκά διαφορετικά ταμεία και τη δίνουμε το λόγο. Ευχαριστώ. Ο στόχος είναι να έχουμε ένα κοινό σύστημα για απλουστευμένους και ενοποιημένους κανόνες για 7 διαφορετικά ε, ταμεία, να μειώσουμε το διοικητικό άχθος ε, για και από τις προγραμματικές αρχές και τους δικαιούχους και να εξασφαλίσουμε την ομαλή ε, εφαρμογή και την τοποίηση των στόχων. Ε, η μακροοικονομική αιρεσιμότητα που προτείνεται, και αυτό το κομμάτι συνδέεται με τη μακροοικονομική αιρεσιμότητα, είναι το πιο σημαντικό τμήμα για την Επιτροπή μας και είναι πολύ παρόμοιο με την ε, τρέχουσα περίοδο, οικονομική περίοδο. Η ευθυγράμμιση των προγραμμάτων πιο στενά με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες και την αυξημένη αποδοτικότητα με πιο στενό σχέση και πιο στενή σχέση με το ευρωπαϊκό εξάμεινο είναι ένα από τους, ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους ε, του κανονισμού. Όμως, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη όμως ότι στην επόμενη περίοδο βάζουμε νέες μετα... Ε, νέα προγράμματα στήριξης των μεταρρυθμίσεων, που είναι στη συνέχεια ε, πιλωτικών προγραμμάτων που είχαμε στην τρέχουσα περίοδο και ο, τρε... ο σκοπός αυτών των προγραμμάτων είναι η εφαρμογή των ειδικών συστάσεων αναχώρα και μια πιο στενή σχέση με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο ο προπολογισμό είναι 25 εκατομμύρια ευρώ για τα προγράμματα στήριξη των επενδύσεων. Ε, το ποσό τη ε, συνοχή ε, στι νέε δημοσιονομικέ προοπτικέ έχει μειωθεί. Στο νέο δεν έχει μειωθεί. Και γι' αυτό νομίζω ότι η πολιτική συνοχή θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο για τι μεταρρυθμίσει. Εάν όλα τα κονδύλια υπό τα προγράμματα στήριξη των επενδύσεων έχουν απορροφθεί και μόνο. Μια άλλη δυσκολία για τι χώρε συνοχή είναι ότι αν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν παράλληλα και τα δύο εργαλεία, δεν θα έχουν αρκετό δυναμικό να το κάνουν. Επομένω, ε, γι' αυτό ακριβώ θα πρέπει να, να, να ε, χρησιμοποιήσουν πρώτα τα προγράμματα στήριξη των μεταρρυθμίσεων. Για τι μεταρρυθμίσει αυτέ καθεαυτέ δηλαδή. Και βεβαίω δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι οι διαφορετικέ μεταρρυθμίσει μπορούν να γίνουν χωρί τουλάχιστον το ίδιο ε, επίπεδο επενδύσεων όπω με την τρέχουσα περίοδο. Ε, γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε νέες θέσεις απασχόλησης, ε, με καλύτερη από παραγωγικότητα, ανταγωνιστικότητα και ποιοτικό επίπεδο. Για την αποτελεσματικότητα των ε, ταμείων και τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση, το Συμβούλιο και η Κομισιόν μπορούν να παίρνουν αποφάσεις χωρίς σαφή θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και μόνο απλώ να μας ενημερώνουν για τα μέτρα και την εφαρμογή των μέτρων. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει όμω. Νομίζω ότι η πρόταση για την αναστολή των, ε, ε, των δεσμεύσεων ή η άρση της αναστολής θα πρέπει να συζητιέται καταρχήν με το Κοινοβούλιο και να υιοθετείται συνεχεία από το Συμβούλιο. Και τέλος, πρέπει να τονίσω ότι καλωσορίζω την εισαγωγή της ρήτρα διαφυγής που επιτρέπει στην Κομισιόν να συστήσει ότι το Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει σε περίπτωση, σε εξαιρετικά ας πούμε, οικονομικά, οικονομικές περιπτώσεις, ε, την αναστολή αυτή ε, ή όταν το ζητήσει με αιτιολογημένη γνώμη το κράτος. Ε, επίσης με τα μέτρα αυτά δεν θα πρέπει να προκαλέσουμε μεγαλύτερη ζημία από όφελος. Πάντα αυτό πρέπει να το μέλημά μας. Ο Ανδρέα Κουτσολίνο από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Καταλαβαίνω ότι καλούμαστε να εξετάσουμε την πολιτική συνοχής και τα εργαλεία της πολιτικής συνοχής με, τα 7, ε, με τους 7 κανονισμούς αυτούς ε, από οικονομική σκοπιά. Πρέπει να τους εξετάσουμε. Πρέπει να υπενθυμίσω όμως και στον εαυτό μου αλλά και στη συνάδελφο ότι εδώ μιλάμε για ένα από τα βασικά εργαλεία που έχει η Ευρώπη στα χέρια της για να μειώσει τις διαφορές, τις αποστάσεις, για να αυξήσει την ανάπτυξη και την απασχόληση των εδαφών μας. Επομένως, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε στην πολιτική συνοχή τα εργαλεία της πολιτικής συνοχής ως μοχλό, ας πούμε, τιμωρητικό απέναντι στα κράτη-μέλη. Επιπλέον, οι πραγματικοί πρωταγωνιστές είναι ε, οι τοπικές αρχές, ε, οι περιφέρειες, ας πούμε, οι κοινότητες, οι δήμοι κτλ. Μην το ξεχνάμε αυτό. Επόμενο, δεύτερο στοιχείο. Η μακροοικονομική αιρεσιμότητα είναι μη εφαρμόσιμη. Όταν προσπαθήσαμε να το κάνουμε, τα καταφέραμε να το κάνουμε. Δεν τα κατάφερε η Κομισιόν, δεν τα κατάφερε το Κοινοβούλιο και επομένω επ' αυτού πρέπει να υπάρχει περαιτέρω προβληματισμό για το θέμα αυτό. Για τη μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Και τέλο, να πω και κάτι άλλο προ τη συνάδελφο. Είχαμε μια συγκεκριμένη εμπειρία. Επαληθεύσαμε πώ η Ελλάδα αυτά τα χρόνια, η οποία δεν χρησιμοποίησε την στη χρηματοδότηση, μπόρεσε να επιταχύνει τη χρήση των ε, κονδυλίων των ταμείων και αυτό ήταν στοιχείο που βοήθησε στην ανάκαμψη. Ε, εγώ πιστεύω ότι μια αύξηση της χρηματοδότησης από πλευρά των ε, κρατών μελών, αν ξεκινήσουμε από εκεί και αν δεν ε, ξαναμιλήσουμε για το ότι αυτό είναι ένα ε, επιπρόσθετο εργαλείο πολιτικής συνοχής και δεν αντικαθιστά την εθνική πολιτική επενδύσεων. Έτσι. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να ξαναπροβληματιστούμε μεταξύ μας. Πώς θα μπορέσουμε προοδευτικά να αξιοποιήσουμε τις χρηματοδότηση και να γίνει αποτελεσματική. Γιατί να μην ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη, στις περιφέρειες, στις αυτόνομες περιοχές, να διπλασιάσουν σε ορισμένε περιπτώσει ω προπόθεση για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τα, τα ευρωπαϊκά ταμεία. Και συνεχεία, αυτά τα κράτη, αυτέ οι περιφέρειες δεσμεύονται πάρα πολύ καλά λόγω του Συμφώνου Σταθερότητα. Τότε στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε την πολιτική συνοχή. Την μπλοκάρουμε αντί να την ε, επιταχύνουμε και να κάνουμε και πιο ποιοτικέ επενδύσει. Επομένω, σα προτείνω κάτι που συζήτηκε πολλές φορές. Πώς θα μπορέσουμε προοδευτικά να ελαφρύνουμε ε, και να αποσυνδέσουμε τη συγχρηματοδότηση από το σύμφωνο σταθερότητα. Αυτά είναι κάποιες ε, ιδέες που θα τις ε, μεταφράσω και σε τροπολογίες. Πιστεύω ότι θα βοηθήσουμε την εισηγήτρια και θα τα δουλέψουμε και στην Επιτροπή Ρέτζι. Από το ECR, ο Στάνισλαβ Όλσο. Ευχαριστώ την Πέρε. που πήρε ότι θα πάρει την Προεδρία για δύο, λόγια, ε, για δύο λεφτά και θα επανέλθω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ συγητή, την Τσίτρια. Η πολιτική μας ομάδα θεωρεί αυτούς τους νέους κανονισμούς που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ σημαντικούς έτσι ώστε πλέον να έχουμε κοινού κανόνε για τα 7 ευρωπαϊκά ταμεία, κάτι το οποίο θα διευκολύνει τη δημόσια διοίκηση των κρατών μελών και επίσης θα καταστήσει τους κανονισμούς αυτούς και πιο ξεκάθαρους. Στις τροπολογίες 1, 2, 5, 6 και 7 υπάρχει αναφορά στην χρήση αυτών των ταμείων για την υποστήριξη των διαρθρωτικών μεταχειριθμίσεων. Όμως αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν είναι γνωστό ακόμα πώς θα λειτουργήσει και γι' αυτό δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Είναι σε αντίθεση με την αρχή του εύνομοθετή το να υποστηρίζουμε τη χρηματοδότηση ενό προγράμματο που δεν ξέρουμε πώ θα εφαρμόστηκε. και ίσω να έρχεται και σε αντίθεση με το εθνικό δίκαιο ορισμένων κρατών μελών. Και Επίσης θα πρέπει να δούμε το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον εποπτικό που θα πρέπει να έχει, του ελέγχου που θα πρέπει να έχει στις τροπολογίες 3 και 11 ε, όσον αφορά τη δυνατότητα να, να αναστέλλεται η χρηματοδότηση, θα θέλαμε να προβλεφθεί και αυτό που ονομάζεται escape clause, η δυνατότητα όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το επιθυμεί να μπορεί να, να υποβάλει την, την έτοιμη, το αίτημα αναστολή στο ε, χρηματοδότηση σε ένα συγκεκριμένο ε, πρόγραμμα στο Συμβούλιο ε, ή με, με κατόπιν αίτημα ε, μέλους πάλι, μέλων. Θεωρούμε ότι σε ορισμένα στοιχεία η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν καλύτερη, ωστόσο βλέπουμε ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποια συμβαστική λύση. Ε, Ραμόν Τρεμόζα για την ΑΛΤΕ. Ευχαριστώ, Περβόνς. Κάθε φορά που συζητάμε το θέμα του πώς αξιοποιούμε τα χρήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι θα πρέπει να γίνεται χρηστή διοίκηση των χρημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζουμε ε, πόσο σημαντικό αυτό είναι. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον, κανονισμό για τις κοινέ προβλέψεις, γιατί αυτό σημαίνει ότι θα είναι πιο αποτελεσματικό και για τις αρχές της ε, ε, εποπτικές και για τις αρχές διαχείρισης. Αυτό θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Το άρθρο 147 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει ότι θα πρέπει να καταπολεμούνται οι διαφορές και οι ανισορροπίες που υπάρχουν μεταξύ των ε, περιφερειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναφερθεί. Η αύξηση της συνοχής μεταξύ των περιφερειών θα πρέπει να είναι ουσιαστικό στοιχείο αυτής της πρόσβασης. Τώρα, για το ζήτημα της αιρεσιμότητας και της σύνδεσης με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Θα θέλουμε περισσότερες ε, διευκρινήσεις για αυτό, γιατί ακόμα περισσότερο δεδομένου ότι θα υπάρξει απλοποιημένη διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις αναχώρα. Στο σχεδιασμό του προγράμματος, στη διάμεση αξιολόγηση και στο κλείσιμο του. Μόνο έτσι μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτές οι συστάσεις θα εφαρμόζονται ουσιαστικά. Σας ευχαριστώ. Euh, merci. Les Verts n'ont pas de représentant. Et donc, je passe la parole au groupe de la GUE. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον Μιγέλ Βιέγκας από την ΚΟΕ. E. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπω. Δυστυχώς ε, δεν συμμερίζομαι την άποψη του εισηγητή, όμως ε, η κριτική μας αφορά τη μείωση ε, των τομέων αρμοδιότητας και τη θεματική συγκέντρωση των διαρθρωτικών ταμείων. Αυτό έχει οδηγήσει Σα ζητώ συγγνώμη, υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη διερμηνία προ τα γαλλικά, λέει η Πρόεδρος. Πράγματι υπήρχαν κάποια περίεργα παράσιτα στο μικρόφωνο. bon, je... Είναι καλά τώρα, μπορώ να ξεκινήσω πάλι. Je ε, Resumindo, não tenho muito a dizer, mas há ακούγεται καλά τώρα η διερμηνία. Ωραία. Λοιπόν, για το ζήτημα της συγκέντρωσης, της θεματικής συγκέντρωσης, για το ζήτημα της σχέσης με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και συγκεκριμένα μιλώντας για την εφαρμογή των συστάσεων αναχώρα σε χώρες τις οποίες υπάρχουν διαρθρωτικές αλλαγές και επίσης όσον αφορά τις μακροοικονομικές, ε, τη μικροοικονομική ερωσιμότητα, θα πρέπει να φροντίσουμε να δίνεται η δυνατότητα σε κάθε κράτος μέλος να εφαρμόζει τις πολιτικές που χρειάζονται για να ανταποκριθεί στις ανάγκες του πληθυσμού ε, και ανάλογα με τις ε, τοπικές ιδιαιτερότητες κάθε περιφέρειας. Γι' αυτόν τον λόγο εμείς έχουμε μια στάση κάπως επικριτική εδώ για τις προτάσεις που βλέπουμε στο τραπέζι και δύσκολα βλέπουμε πώς θα μπορέσουμε να, ε, να καταλήξουμε σε συμβιβασμό. Θα υποβάλουμε παρόλα αυτά τις τρο, ε, τροπολογίες μας με την ξεχωριστή δική μας θέση, λέγοντας καταρχήν ότι η θέση μας επί τους πρότασης που βλέπουμε είναι αρνητική. Η Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Θα ρωτήσω αν υπάρχει κάποιος άλλος συνάδελφος που ζητά το λόγο. Όχι από ό,τι βλέπω. Κυρία Μάλετιτς, μήπως θέλετε να Λάβετε το λόγο για να δευτερολογήσετε. Κυρία Μαλέτιτς, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους σκιώδει εισηγητέ. Συμφωνούμε όλοι ότι στόχος δεν είναι να τιμωρηθεί κάποιος από τους δικαιούχους, αλλά να υπάρχει καλύτερη επίτευξη των στόχων της περιφερειακής πολιτικής, των μακροοικονομικών στόχων. Γι' αυτό το λόγο κανείς θα πρέπει να είναι ε, προσεκτικός στην εφαρμογή αυτών των μέτρων για να μην δημιουργήσει μεγαλύτερη ζημιά από τι όφελο. Γι' αυτό το λόγο ο συνάδελφος λέει ότι δεν είναι σωστό να αναφερθούμε στην πρόταση για την ε, υποστήριξη των προγραμμάτων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, μιας και η Κομισιόν δεν έχει υποβάλει ακόμα τη σχετική πρόταση. Όμως, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να τα δούμε το θέμα αυτό και το θέμα αυτού του, του, της, της πρότασης από κοινού. Είναι ένα πακέτο. Έχει υποβληθεί τροπολογία για να διαγραφεί η σχετική πρόβλεψη. Όμως, στόχος δεν είναι να σταματήσει η εφαρμογή της περιφερειακής πολιτικής, στόχος είναι να βελτιωθεί η υλοποίηση των συστάσεων αναχώρα. και γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει τροπολογία για τη διαγραφή. σα. ευχαριστώ. Και εμεί σα ευχαριστούμε να σα υπενθυμίσουμε το ε, χρονοδιάγραμμα. Προθεσμία για τις ε, τροπολογίες 9 Οκτωβρίου, 12 η ώρα. Ξέδεση τροπολογιών 12 Νοεμβρίου. Την ίδια ημέρα ψηφοφορία στην ε, ΕΚΟΝ. Η Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής ΡΕΤΖΙ θα ψηφίσει στις 3 Δεκεμβρίου. Προχωρούμε με την ημερήσια μας διάταξη και πρόκειται για τη γνωμοδότηση την οποία θα ε, υποβάλουμε στην ΑΦΚΟ, είναι η έκθεση Φρουντσούλιτσα για την διαφοροποιημένη ενοποίηση. Το φαινόμενο αυτό της μεταβλητής ολοκλήρωσης δεν είναι καινούριο είναι κάτι το οποίο το συζητούμε από τη δεκαετία του 70 και εντάθηκε η σχετική συζήτηση το 90. Θα σας δώσω ορισμένα παραδείγματα. Η δυνατότητα, η δημιουργία μάλλον της ΟΝΕ το 1993. Είναι ένα παράδειγμα ολοκλήρωσης με διαφορετικό ρυθμό. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ένα εργαλείο για να, να υπάρχει ολοκλήρωση προσαρμοσμένη στις ε, πολιτικές πραγματικότητες. Όμως θα πρέπει να γίνει με τρόπο ε, πιο ε, λογικό και με μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμοποίηση. Αυτή η διαφοροποιημένη ολοκλήρωση φαίνεται ιδίω στι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που πρόσφατα ήρθαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργεί την εντύπωση ότι είναι εργαλείο για να δημιουργούνται πολλέ ταχύτητε. Στην πραγματικότητα, η... έχουν αυξηθεί οι διάφορες πολιτικές τις οποίες υλοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και η γενικότερη της εμπάθυνση και ολοκλήρωση. Πρόκειται για έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, η οποία αφορά ουσιαστικά τη θεσμική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως είναι σημαντικό να καταγράψουμε και εμείς μια ενθάρρυνση προς το μοντέλο opt-in προς τα κράτη-μέλη. Όποιο μοντέλο και αν τελικά γίνει δεκτό ε, στο μέλλον για την οικονομική ολοκληρώση. συμφωνούμε όλοι στο εξή ότι όταν υπάρχουν διακρατικές διαδικασίες, αυτό ε, ε, οδηγούμαστε σε πιο περίπλοκες διαδικασίες και με μικρότερη δυνατότητα δημοκρατικού ελέγχου. Η κοινοτική μέθοδος, που είναι δυναμική όχι στατική, είναι κατά την άποψή μου ο καλύτερος τρόπος λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως η κοινωνική μέθοδος θα πρέπει να ανανεωθεί και να χρησιμοποιείται περισσότερο. Μεταξύ όλων αυτών των στόχων λοιπόν, αναφέρω τη σημασία που έχει να ενισχυθεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων και στην οικονομική διακυβέρνηση, έτσι ώστε να ενισχυθεί ο δημοκρατικός έλεγχος και των διατάξεων για την ε, οικονομική διακυβέρνηση ε, και με πλήρη σεβασμό στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους τομείς αυτούς. Το Brexit μας δίνει τη δυνατότητα να απομακρυνθούμε από το μοντέλο opt-in, opt-out προς ένα περισσότερο μοντέλο, περισσότερη, μεγαλύτερη χρήση ενός μοντέλου opt-in, το οποίο στην πραγματικότητα θα δώσει ευελιξία και θα ανοίξει την πόρτα στις χώρες εκείνες του που το επιθυμούν και πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια να προχωρήσουν όσο γρήγορα χρειάζεται. Επίσης θα ήθελα να τονίσω τη σημασία που έχει η χρήση των διαρθρωτικών ταμείων, του, ταμείου, του Ταμείου Συνοχής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ταυτόχρονα. και να καλωσορίσουν και τα νέα προγράμματα τα οποία προγραμματίζονται, όπω για παράδειγμα τα προγράμματα ενίσχυση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για εκείνε τι χώρε οι οποίε πρόκειται και προσπαθούν να μπουν στο ευρώ. Θα χρειαστεί ε, να αυξηθεί ο προπολογισμό που η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει σε τέτοια προγράμματα. Με χαρά θα συνεργαστώ με τους συναδέλφους Σκιώδης και με χαρά θα περιμένω τις τροπολογίες σας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν είναι εδώ όλοι και όλοι οι συζητητές. Από τους φιλελεύθερους. Α, θα πάρει το λόγο ο ξενόματος του ΕΛΚΑ. Η κυρία Μάλετιτς. Που θα αντικαταστήσει τον Αλά Λαματσού. Ευχαριστώ. Γκάλαν Λαμασούρ prepared uh, uh Λαμασούρ ετοίμασε κάποια σημεία, θα τα διαβάσω έχει το σχέδιο γνωμοδότηση διάφορε ενδιαφέρουσε παρατηρίε για του μηχανισμού ε, τη ρήτρα προσχώρηση για να επανεστιάσει η συζήτηση στην ενδοενωσιακή ολοκλήρωση παρά στι σχέσει με τρίτε χώρε. Η παράγραφος για την ε, ολοκλήρωση της, ε, του μηχανισμού σταθερότητας στις συνθήκες είναι εκτός θέματος. Σε ό,τι αφορά την τελευταία παράγραφος, η έμφαση θα πρέπει να δοθεί σε πολιτικές οι οποίες δίνουν κίνητρα για την ολοκλήρωση. Όλες αυτές που αναφέρθηκαν θα πρέπει να είναι προσπελάσιμες σε όλες τις ευρωπαϊκές ενωσιακές χώρες. Δεν έχει κανένα νόημα να τις αναφέρουμε ε, λοιπόν σε μια έκθεση για τη μεταβλητή ολοκλήρωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και μια και δεν υπάρχει εκπρόσωπος του ECR, Θέλετε να πάρετε το λόγο. Α, με συγχωρείτε. Δεν σα είδα να φτα... καταφθάνετε, κύριε Σταρμπάτη. Ναι, ναι, συγγνώμη, κοίταξα το χρονοδιάγραμμα τη ημερήσια διάταξη και μπερδεύτηκα. Ναι, ναι, έχω κάποια σχόλια να κάνω για τι προτάσει που βλέπουμε εδώ. Το βλέπω από άλλη οπτική γωνία. Η διακυβερνητική διαδικασία βεβαίως και θα συνεισφέρει στην ε, μείωση της ε, διαφάνειας και θα υποσκάψει ε, τις προσπάθειες. Αυτό για μένα είναι σαφές. Το βλέπουμε. Βλέπουμε και αυτά που είπαν και ο Μοσκοβισή και ο Μακρόν για την ε, περίπτωση της Ελλάδας. Περισσότερος δημοκρατικός έλεγχος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακούμε. Αυτό για μένα είναι ενίσχυση της, ε, του συγκεντρωτισμού. Ε, η ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, η αύξηση των αρμοδιοτήτων του έναντι των κρατών μελών, έναντι της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, έναντι των εθνικών κυβερνήσεων. Αυτό είναι μια ισοπαίδωση. Αυτό μην ξεχνάτε, το ανέφερε και ο Υπουργό Οικονομικών κ. Σόλτ. Ε, Η πρόταση του σημείου 2 δεν είναι τίποτα άλλο από μία προσπάθεια συγκεντρωτική για ε, κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε αύξηση της ε, γραφειοκρατίας, να είστε σίγουροι. Αυτό είναι δημοκρατικός συγκεντρωτισμός, αν θέλετε. Σημείο 5. Εδώ νομίζω πως προσπαθούμε να κάνουμε το κατόρθωτο. Βλέπουμε ότι όμως αυτές οι προσπάθειες είναι κάπως υπερβολικές. Ε, δεν θεωρώ πως αυτό οδηγεί στην ε, ολοκλήρωση. Δεν θεωρώ πως μακροπρόθεσμα θα έχει και νόημα να διαθέτουμε χρηματοδοτικά κονδύλια τα οποία δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε δεν βλέπω μεταβλητή ολοκλήρωση με αυτήν την έννοια. Αντιθέτως, ε, αυτή η έκθεση που βλέπω είναι μια έκθεση για την αύξηση του συγκεντρωτισμού στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που τηρήσατε και το χρονο, χρονικό όριο. Και τώρα, κυρία Λίβερινγκ από τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Φρουτζουλίτσα, αγαπητοί συνάδελφοι, καλωσορίζω το σχέδιο έκθεσης, διότι είναι σαφές, σύντομο και περιγράφει με ακρίβεια το πώς θα προχωρήσουμε. Είναι μια ενωσιακή μέθοδος που θα ορίσει το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διακυβερνητικές δομές είναι χρήσιμες όταν ε, έχουν νόημα, όμως βλάπτουν όταν ε, παρεμβαίνουν σε αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, διότι μόνο η Ένωση μπορεί να ε, δώσει λύσεις τόσο ευρείες. Μπορούμε να συζητήσουμε βέβαια πολλές από αυτές τις ε, προτάσεις, μπορούμε να συζητήσουμε το πλαίσιο. Για μένα βέβαια η έμφαση θα πρέπει να δοθεί σε μια ισχυρότερη οικονομική και νομισματική ένωση. Κάποια σχόλια τώρα. Η ευθύνη πρέπει να συνοδεύεται και από λογοδοσία. Αγαπητοί συνάδελφοι, μία ολοκληρωμένη ένωση δεν είναι μία ένωση ε, μεταφορών κεφαλαίων. Έπειτα, η θεσμοθέτηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, σταθερότητας παρά το ότι είναι ε, καλό μου με παραπέμπει σε ένα μεγαλύτερο πρόβλημα. Πώς μπορούμε δηλαδή ε, να κάνουμε κάτι τέτοιο εάν δεν συμμετέχουν όλοι σε μια πολιτική η οποία δεν χρηματοδοτεί επίσης όλους. Η ολοκλήρωση χρειάζεται χρόνο. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει τουλάχιστον να υπάρχει ένας ε, οδικός χάρτης που ε, να δίνει με σαφήνεια την ε, κατεύθυνση. Ολοκλήρωση, ναι. Όμως Ευρώπη Αλακάρτ, όχι πλέον. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Βιέγας. Θέλετε να εκπροσωπήσετε την ΚΟΕ, μια και ο σκιώδης συγκητής δεν είναι παρόν. Όχι. Τότε ξαναδίνω το λόγο στον κύριο Φρουντσούλικα. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που παρενέβησαν για αυτό το θέμα. Πρέπει να συνεργαστούμε. Καταλαβαίνω τις θέσεις σας. Και φυσικά είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να έχουμε όλες αυτές τις συμφωνίες για, τις, συμφωνίες για την ε, Οικονομική και Νομισματική Ένωση για όλα τα, ε, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέλλον τη στιγμή που θα είναι έτοιμα για να υιοθετήσουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ούτως ώστε να μπουν στην Ευρωζώνη και στην ε, Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση. Παράλληλα, η κατάσταση δεν είναι εύκολη, γιατί διάφορες ισχυρές φωνές ε, από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη λένε ότι πρέπει να προχωρήσουμε, αν γίνεται, όλοι μαζί. Ότι δεν πρέπει να δημιουργούμε δεν πρέπει να δημιουργούμε ρήγματα ανάμεσα στην Δυτική Ευρώπη, ας πούμε, μια ένωση των δυτικών ευρωπαϊκών χωρών και των ανατολικών χωρών. Θα πρέπει όλες οι χώρες μέλη της Ένωσης που το ζητούν να είναι μέλος της Οικονομικής και Νοσηματικής Ένωσης και να αφήσουμε την πόρτα ανοιχτή στο μέλλον για όλες τις χώρες μέλη που θέλουν να ενταχθούν. Να μπουν στην ΟΝΕ. Επίση, μην ξεχνάμε και τι χώρε που θα ενταχθούν στο μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό να σταματήσουν όλε αυτέ οι ρήτρε προσχώρηση και αυτοεξαίρεση. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα, το πρόβλημα είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τι χώρε που είναι ήδη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε χώρε με 4 opt-out ή 5 opt-out, ας πούμε. Δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιες ρήτρε να έχουμε μέλη, να έχουμε χώρες οι οποίες, όπως είπε και ο συνάδελφος εδώ, ε, ή συνάδελφος μάλλον, ότι επιλέγουν τα καλά και πετάνε ότι τους αρέσει. Δηλαδή μια Ευρώπη αλλά la carte. Δεν γίνεται. δεν μπορούν να υποφελούνται μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να πετούν τα υπόλοιπα που δεν του αρέσουν. Νομίζω ότι θα πρέπει να σταματήσουν αυτέ οι ρητρε opt opt-in και opt-out. Όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δεχτούν την Ένωση ω έχει, συνολικά. Και θα πρέπει να σταματήσουν οι ρήτρε αυτοεξαίρεση επί διαφόρων θεμάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σιγητά. Πολύ ωραία. Ε, για τις τροπολογίες, 9 ε, Οκτωβρίου στις 12 είναι η προθεσμία. Ε, η εξέταση και η ψηφοφορία θα γίνει στις 12 Οκτωβρίου, όχι στις 12 ε, Νοεμβρίου, διορθώνει ομιλήτρια. Θα ψηφίσουμε στην ΑΦΚΟ κάποια στιγμή μετά, φυσικά. Πολύ ωραία. Πάμε στο σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης. Πρόκειται για την αρμόνιση των ε, διαρθρώσεων των φόρων κατανάλωσης στο τομέα της αλκοόλης, της αλκοόλης και των αλκοολούχων ποτών. Και ο εισηγητής μας είναι ο Μιγγέλ Βιέγας. Έχει το λόγο. Ε, Σας ευχαριστώ, θα είμαι σύντομος. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία χρήσιμη. Το θέμα για το οποίο συζητούμε είναι ένα ζήτημα στο οποίο διαπιστώνουμε ότι υπάρχει διαφορετική ερμηνεία και άρα διαφορετική εφαρμογή των κανόνων για, τα ειδικά, για τους ειδικού φόρους κατανάλωσης όσον αφορά τα αλκοολούχα ποτά από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Και με αυτόν τον τρόπο, ε, με αυτήν, η πρόταση μάλλον προσπαθεί να λύσει αυτό το πρόβλημα και να υπάρξει εναρμόνιση στις ε, εξαιρέσεις που υπάρχουν είτε για την καθαρή αλκοόλη καθώς επίσης και για τα αλκοολούχα ποτά ε, όπως αυτά ε, σιγά σιγά εμφανίζονται. Ε, γιατί υπήρξε μια κατάσταση στην οποία τα ο ειδικό φόρο κατανάλωση δεν εφαρμοζόταν με τρόπο ενιαίο. Και ο τρόπος με τον οποίο επιδιώκει αυτό τον στόχο η πρόταση είναι τέτοιος που δεν θα δημιουργήσει προβλήματα στους εμπορευόμενους, τους επιχειρήσεις του κλάδου, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι τεχνικό και περίπλοκο. Η πρωτοβουλία όμως είναι απολύτως απαραίτητη. Και σε αυτό το πνεύμα συνέταξα και την έκθεση την οποία έχετε στα χέρια σας. Βεβαίως θα ακούσω τις παρατηρήσεις που θα κάνετε στο προσχέδιο της εκθέσης μου. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για το ΕΛΚ. Ο κύριος Ντόρφμαν. Ευχαριστώ. Συμφωνώ πλήρως με τον, με τον εισηγητή, με την έκθεση. Είναι πράγματι τεχνικού χαρακτήρα και προσπαθεί να λύσει κάποιες προβλήματα που υπήρχαν στην ερμηνεία των ειδικών φόρων για τα αλκοολούχα. Για, στο άρθρο 1 και συγκεκριμένα στην πρώτη τροπολογία θα ήθελα να μου διευκρινιστεί τι προβλέπετε για τη σύνθεση της μπύρας. Πώς θα γίνονται οι μετρήσεις συγκεκριμένα των σακχάρων με ποια μεθοδολογία δεν είναι πολύ ξεκάθαρο για εμένα αυτό μονάχα. Κατά τα άλλα, θα έλεγα ότι η πρόταση είναι ουσιαστική. Κατάλαβα όμως ότι θα ήθελα να επισημάνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει καταφέρει να μας υποβάλει μία πρόταση η οποία να είναι ουσιαστική και να ρυθμίζει το ζήτημα των ειδικών φόρων κατανάλωσης για τις πωλήσει αλκοολούχων ποτών online μέσω ίντερνετ. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο φέσταται εδώ και πολύ καιρό και δημιουργεί ε, σημαντικό διοικητικό άχθος σε όλα τα κράτη-μέλη. Αυτές οι πωλήσει στο ίντερνετ των αλκοολούχων ποτών. Δημιουργείται σημαντικό διοικητικό άχθος. Και πώς και δεν καταφέρνουμε να λύσουμε το ζήτημα αυτό, να έχουμε μια ουσιαστική πρόταση για το θέμα αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μια πρόταση που να είναι υπέρ του ε, καταναλωτή. Είναι απίστευτο ε, να έχω τη δυνατότητα να πάω σε ένα άλλο κράτο μέλο, να γεμίσω το πόρμπαγκάζ μου με αλκοόλ και να γυρίζω σπίτι. Όμω, ε, όταν θέλω να αγοράσω ένα μπουκάλι ε, ποτό από το ίντερνετ, να μην γίνεται αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματικά μετά από πάρα πολλά χρόνια υπέβαλε μία λογική κατά με πρόταση για να λύσει αυτό το πρόβλημα και να ε, μην ε, πληρώνει τα σπασμένα ο ε, καταναλωτής. Σας ευχαριστώ. Πολύ ωραία. για την πύρα μιλάμε. Πολύ ιδιαίτερα ειδικά σημεία από τους σοσιαλιστές. Σας ευχαριστώ πολύ. Οι σοσιαλιστές και δημοκράτες συμφωνούν με τον ε, εισηγητή κύριο Βιέγας. Στηρίζουμε την πρόταση της Επιτροπής και θεωρούμε πως η ρύθμιση αυτή για ε, τον φόρο κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών πρέπει επιτέλους να αλλάξει. Η δυνατότητα όμως ε, και οι ευκαιρίες που μας δίνει η τεχνολογία πρέπει να χρησιμοποιηθεί, πρέπει να αξιοποιηθεί ζητούν ε, διοικητικές διαδικασίες οι οποίες δυσκολεύουν τη ζωή των ε, παραγωγών, των ε, μεταπολιτών να διαθέσουν τα προϊόντα. Αυτό γίνεται εις βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θεωρώ πως ε, θα πρέπει για τους μικρούς ε, παραγωγούς να, υπάρχει, να υπάρχουν λογικοί φορολογικοί συντελεστές ή συγκεκριμένες διατάξεις που ε, να ρυθμίζουν ειδικέ μπύρες, για παράδειγμα αρωματικές μπύρες, μπύρες με γλυκαντικές ουσίες. Πρέπει να γίνει μια διαφοροποίηση. Γι' αυτό λοιπόν καλωσορίζω την έκθεση του εισηγητή. από τους φιλελεύθερους ο κύριος ε, Ραμόν Τραμόζα. Ευχαριστώ. Μιλάμε για απλουστευμένη διαδικασία. Ε, υποστηρίζει ο εισηγητή την πρόταση τη Κομισιόν και εμεί ε, επίση ε, την υποστηρίζουμε, όπω είπαν και όλοι οι προλαλήσαντε. Έχουμε κάποιε ανησυχίε όμω ε, που μας έχουν διαμηνήσει κάποιοι μικρή παραγωγή, οικογενειακή, κάποιε επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν, α πούμε, πριν από 100 χρόνια στη δική μου εκλογική περιφέρεια, αλλά και αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητούμε να, να καλύψουμε τα τρόφιμα και τα ποτά με πιο ισορροπημένο τρόπο. Ε, τα κίνητρα για τους μικρούς ε, παραγωγούς είναι ότι ε, θα πρέπει να έχουν μειωμένους συντελεστέ. Θα πρέπει να ξέρουν ότι οι μειωμένοι συντελεστές ε, αφορούν όλα τα ποτά, ε, την πύρα, το, το κρασί κτλ. Αν η οδηγία έχει ε, διαφορετικές, ε, διαφορετικές προϋποθέσεις για τους μειωμένους συντελεστές από ότι για τους άλλους συντελεστές, ας πούμε, θα έχουμε ε, μεταχείριση των μικρών παραγωγών, των μικρών ιστοποιών κτλ. σε σχέση με τους άλλους. και η ανισορροπία θα επιταθεί. Αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, ζητούν λοιπόν μεγαλύτερη δικαιοσύνη, ούτω ώστε ε, να έχουν τις ίδιε φορολογικέ προτιμήσει, ε, μάλλον τις ίδιες, τη ίδια φορολογική μεταχείριση μικρή παραγωγή με του μεσαίου ε, παραγωγού. Επίσης, πρέπει να ξαναδούμε και τους ειδικού φόρους κατανάλωσης. Ε, για, μιλάμε για ποτά που έχουν χαμηλό αλκοολικό τίτλο. Ε, la question, Η Βερνιά δεν είναι εδώ. Ποιος θα υποστηρίξει τον εισηγητή, δηλαδή να πάμε προς μια προστευμένη νομοθετική διαδικασία, δηλαδή χωρίς τροπολογίες. Είναι μια πρόταση η οποία θα μπορούσε να γίνει δεκτή από όλους. Έχουμε την πρόταση Κομισιόν δηλαδή και με την απλουστευμένη διαδικασία να προχωρήσουμε. Ναι, δεν υπάρχουν ιδιαίτερε αντιρρήσει. Πολύ ωραία. Θα προχωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Και επομένω, τι σημαίνει αυτό. Θα ακολουθήσουμε τον κανόνα, τον, ε, το άρθρο 51 μάλλον. Άρθρο 51. Και ψάχνω λίγο τα γαλλικά μου. Και άρα μπορούμε να προγραμματίσουμε την έκθεση του κυρίου Μιγγέλ Βιέγα για να ψηφίσουμε κατευθείαν στα Λομέλια. Υπάρχουν άλλα σημεία που θα θέλατε να θέσετε. Όχι. Και επομένω, τελειώσαμε εδώ. Εποφελθείτε από το βράδυ στο Στρασβούργο. Γεια σας.